Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Προτείνω να ξεκινήσουμε γιατί χθε κατά τη διάρκεια τη απογευματινή συνεδρία υπήρξε ένα θέμα τη ημερησία διάταξη το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε. Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ Ευρωπαϊκή Ένωση επέκεινα του 2020. Προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε πρώτα αυτό το θέμα και μετά τα υπόλοιπα θέματα τη ημερησία διάταξη ω είχαν αναφερθεί, που είναι τα θέματα των ε, τρίτων ε, υπηκών τρίτων χωρών που έχουν βίζα όταν διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Παίρναμε λοιπόν πρώτα στο σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Κόουσο Περμούι για το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και επέκεινα του 2020. Σας υπενθυμίζω ότι η Συμφωνία του Κοτονού θα εκπνεύσει το 2020. Από το 2000 η Συμφωνία της Κοτονού είναι η βάση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 79 χώρες ΑΚΕ και περιλαμβάνει πολιτικό διάλογο, ανάπτυξη και εμπόριο. Επειδή αλλάζει το παγκόσμιο πλαίσιο και υπάρχουν νέε θεσμικέ, πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι χώρε ΑΚΕ, θα πρέπει να σκεφτούμε αν το πλαίσιο αυτό είναι ακόμα έφορο την τωρινή του μορφή και τι αλλαγέ πρέπει να γίνουν. Οι συζητήσει για την συνέχεια τη Κοτονού έχουν ήδη ξεκινήσει και θα υπάρχουν σημαντικέ συνέπειε και για τι χώρε ΑΚΕ αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξωτερική τη δράση. Με την γνωμοδότησή μα, εμεί θα συμβάλλουμε σε μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Ο κύριο Κόουσο ζήτησε συγγνώμη διότι δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Λόζιν, η οποία θα παρουσιάσει αυτή τη γνωμοδότηση εξ του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ο κύριος Κόουσο δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα γιατί έχει σημαντικές ε, ε, υποθέσεις στην Ισπανία. Σας ζητά και πάλι την επίκεια και την κατανόησή σας. Η γνωμοδότηση αυτή έχει σαν στόχο να εξετάσει την συνέχεια των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ και να τις θέσει σε μια νέα βάση. Μια βάση που να έχει ισότητα μεταξύ των δύο εταίρων και να βασίζεται στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει οι εταίροι αυτοί να επιδιώξουν την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της χιλιετίας και να ασχοληθούν με τα θέματα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι αρνητικές συνέπειες των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και σύνδεσης με τις χώρες ΑΚΕ είναι φανερές. Γι' αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό να μπορέσουμε να σκεφτούμε για μια νέα μορφή διάρθρωσης αυτής της εταιρικής σχέσης και οι δικές μου προσωπικές απόψεις είναι κάτι που έχει αναφερθεί και είναι και δική μου άποψη, λέει ο κ. Κόβους, αλλά είναι και πράγματα που έχει τονίσει και ο πρόεδρος μας, ο κ. Μπρόκ, σε συνεντεύξεις με γερμανικά έντυπα και τηλεοράσεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν στο πλαίσιο αυτό να εξασφαλίσουμε την προστασία της γεωργίας, να αντιμετωπίσουμε την υπερβολική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, αλλά και την αρπαγή γης και να διατηρήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες αυτές. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η νέο απικιακή πολιτική που ασκείται μέσες φορές κατά των χωρών ΑΚΕ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να σταματήσουν και οι παρουσίες ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στις χώρες ΑΚΕ. Εμείς ακολουθούμε λοιπόν την γραμμή των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρξει ένα κράτος δικαίου με τις απαραίτητες υπηρεσίες προς τους ανθρώπους. Θα πρέπει οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των ανθρώπων στις χώρες αυτές, να μην υπάρχει νέα μορφή δουλείας, να μην υπάρχουν παράνομες ροές μαύρου χρήματος και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα υποστηρίζουμε, όπως και την αναδιάρθρωση των κρατικών ε, χρεών και την αίτηση των χωρών ΑΚΕ να ελεγχθούν και πάλι τα χρέη τους και να υπάρξει ελάφρυνση αυτού του χρέους. Επίσης πρέπει να υπάρξει αποσημείωση των χωρών ΑΚΕ λόγω της καταλήστευσης των φυσικών σπόρων από ξένες επιχειρήσεις και τις ε, πολεμικές ενέργειες που έχουν προωθήσει αυτές οι πολυεθνικές εταιρείε. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει δικαιοσύνη και ισότητα μεταξύ χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα πρέπει να σκεφτόμαστε τους λαού αυτών των χωρών και όχι μονάχα του αιματοβαμένου ολιγάρχε. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος, κυρία Λέζινγκ. Τώρα, να δώσουμε στον συντονιστή του κύριο το λόγο για το ΕΛΚ, ε, γιατί η ισχύωση δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Πρέντα. Ναι, ναι, όντω η κυρία Μαρία Γκαμπριέλ που είναι η δική μα ε, συγκέντρια δεν παρίσταται, αλλά έχει αποστείλει ένα σημείωμα με την άποψή τη το οποίο και σα διαβάζω. Και λέει ότι το σχέδιο κειμένου ε, πάσχει, είναι ε, λοιπέ, είναι ιδεολογικά φορτισμένο όσον αφορά τις σχέσεις με το 2020 και όπως είναι τα πράγματα τώρα εμεί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κείμενο. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε το ότι θα πρέπει να τονιστεί τεμένη αξία από μια εταιρική σχέση και θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή και αναβαθμισμένη η κοινοβουλευτική διάσταση. Οπότε κάνει τη σχέση εδώ με τη σύνδεση η κυρία Γιαβριέλ με μια πρόσφατη γνωμοδότηση ε, στην Επιτροπή Ανάπτυξης και αφορά την συνοχή ε, των πολιτικών μας ε, που πρέπει να εξυπηρετούν την ανάπτυξη ακριβώς όπως ειδήθηκε στο Στρασβούργο. Προσθέτει κύριε Γκαμπριέλ ότι θα πρέπει να πετύχουμε τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη 2030 και θα πρέπει επομένω αυτά να γίνουν στα πλαίσια των σχέσεων ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2030 για πολιτική συνεργασία πρέπει να τύχει ανανέωσης και είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αναφέρει η κυρία Γκαμπρίελ, να μιλήσουμε και για την πτυχή της ανάπτυξης για την ε, ασφάλεια και ε, θα πρέπει επομένως να έχουμε το African Peace Facility το οποίο ίσχυε και θα πρέπει να προβληματιστούμε τι θα το διαδεχθεί γιατί αυτή τη στιγμή δεν φύγει το ζήτημα αυτό στο σχέδιο κειμένου. Και η συγγήτρια για το ΕΛΚ θεωρεί ότι λείπει από το κείμενο του κ. Περμούη ο αυθεντικός προβληματισμός για έναν πολιτικό διάλογο. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη, ο πολιτικός διάλογος δηλαδή, δυνάμη των άρθρων 8 και 96 και σε τρεις αυτές περιφέρειες και να υπάρξει μια διαδικασία αναθεώρησης, ούτως ώστε να γίνει ανανέωση της σχετικής συνθήκης. Αυτά για το ΕΛΤ. Ευχαριστούμε Κριστιαν, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα να δώσουμε τον ε, λόγο στον συνάδελφο Ζάλα γιατί είναι ο σκιώδης ηγητής για τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Συνάδελφοι, λέει ο κύριος Ζάλα, ο εισηγητής, είχε φιλοδοξίες προετοιμάζοντας το σχετικό κείμενο. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι ο ρόλος της ε, ΑΦΕΤ είναι όχι το να προβάλλει την διεθνή συγκυρία, αλλά να προβάλλει τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της εκθέσεις. Να, πώς μπορεί να έχει προσθέμενη αξία δουλειά της Επιτροπής μας. Ας μην ξεχνούμε ότι οι αναπτυξιακές εμπορικές συναλλαγές καλύπτονται ή θα έπρεπε να καλύπτονται από το σχέδιο κειμένου της Επιτροπής Ανάπτυξης. Εμείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα στρατηγικά μας συμφέροντα στις σχέσεις μας με τις χώρες ΑΚΕ. Η αναβάθμιση δηλαδή της ε, πολυμερούς πτυχής της λειτουργίας αυτής της ε, σχέσης και σε πολιτικό επίπεδο η έκθεση αυτή απλώς επικρίνει το, την νεοαπικία απεικιοκρατική συγγνώμη, πολιτική. Εμείς γιατί έχουμε κατεβάσει κάποιες τροπολογίες ως σοσιαλδημοκράτες. Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί τελικά ε, κάποιος ε, άρτιος συμβιβασμός για να οδηγηθούμε σε μια αξιολόγη έκθεση. Ευχαριστούμε συνάδελφε Ζάλα, λέει ο Πρόεδρος. Από ό,τι βλέπω δεν έχει άλλο τον ε, λόγο. Άλλωστε λείπουν και κάποιοι των σχεδόν συγκεκριτών. Α, η κυρία Θεοχάρου είναι εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και τα ζητήματα ασφάλειας ε, όπως και το μεταναστευτικό το οποίο είναι ένας ισχυρός αποσταθεροποιητικός παράγοντας καλές διμερείς σχέσεις, η απαλλαγή από τις νέο-απικιακές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν κάποια κράτη ή κάποιοι παράγοντες, για να μην το προσδιορίσουμε μόνο σε επίπεδο κρατών, και, και κυρίως η πολιτική ασφάλειας δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν παρά μόνο με την ανάπτυξη των ε, χωρών ΑΚΕ και η ανάπτυξη δεν μπορεί να ξεκινήσει παρόλο που έχει τονιστεί πολλές φορές στις ε, εκθέσεις της Επιτροπής ΑΦΕΤ ούτε μέσα της ε, ΔΕΒΕ ούτε μέσα από πολυδάπανους πολιτικούς διαλόγους και συχνές συναντήσεις αλλά με την στόχευση κυρίως στις κοινότητες των χωρών αυτών και την παράκαμψη των διεφθαρμένων ως συνήθως κεντρικών κυβερνήσεων. Εμείς επιμένουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα παιδείας, δηλαδή η απάντηση είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της παιδείας, της μεταφοράς ε, ικανοτήτων και γνώσεων τα ε, κατοίκους των χωρών αυτών, αφού αντιμετωπιστεί πρώτα το οξύ πρόβλημα της πείνας, της φτώχειας και στοιχειοδός η ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας με την ενίσχυση κυρίως των περιφερειακών ε, ε, περιοχών της, ε, των χωρών αυτών. Ε, αυτά έχουν καταγραφεί σε πάρα πολλές εκθέσεις και της ε, ΔΕΒΕ και σε, ε, της Μιχτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και νομίζω ότι η επανάληψή τους χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα δεν δίνει ε, καμιά βοήθεια προς τις χώρες ΑΚΕΣ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Θεοχάρους. Νομίζω ότι έτσι εξαντλήσαμε τουλάχιστον ε, τα αιτήματα για να πάρετε το λόγο. Η κυρία Λούση νομίζω πολύ καλά παρουσίασε τα θέματα που τίθενται στο σχέδιο. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο. Συνεπώς όσοι θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες ώστε να τα λάβει υπόψη τη ΣΥΝΤΕΒΕ μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ωραία, και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη και συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στις εξαιρέσεις όσον αφορά τις θεωρήσεις, αυτή τη φορά για την Ουκρανία. Και χτες συζητήσαμε, συζητήσαμε μια αντίστοιχη πρόταση όσον αφορά την Γεωργία. Η εισηγητής μας για την γνωμοδότηση αυτή είναι ο συνάδελφος Σάριους Βόλσκι που είναι ο μόνιμος εισηγητής για την Ουκρανία. Γνωρίζετε ότι το θέμα ε, της κατάργησης ε, των θεωρήσεων, ε, ο διάλογος ο σχετικό έχει αρχίσει από το 2012 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει πρόσφατα σχετική έκθεση και η πρόταση όσον αφορά την Ουκρανία ήρθε μετά από μια πολύ σε βάθος αξιολόγηση των απαιτήσεων και των προγραμμάτων δράσης όσον αφορά ε, τα προαπαιτούμενα για την κατάργηση των θεωρήσεων. Τα πράγματα είναι τώρα σε επίπεδο Κορεπέρ και Συμβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό και εμείς ως Κοινοβούλιο να διαρθρώσουμε την ε, συζήτηση βασιζόμενη στις ε, ικανότητες και στα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας χωριστά. Η Μαρία Κάμπριελ είναι η συγγήτρια για τα θέματα αυτά και σίγουρα το Κοινοβούλιο πρέπει να δράσει γρήγορα και οι λόγοι γι' αυτό να υπάρχουν βέβαια και στην αιτιολογική σκέψη που υποβάλλει ο κύριος Άριος Βόλσκι. Όποιος θέλει το λόγο για αυτό το θέμα παρακαλώ να με ειδοποιήσει. Αλλά πρώτα ο εισηγητής μας, ο κύριος Σάριος Βόλσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να ασχοληθεί με το θέμα αυτό της κατάργησης των θεωρήσεων. Είναι σαφές ότι πρόκειται για θέμα εξωτερικών υποθέσεων. Οπότε έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά συγχρόνως θα κάνω έκκληση στην ηγεσία της Επιτροπής μας, Πρόεδρε. Λέω ότι κάνω έκκληση στην ηγεσία τη Επιτροπής μας, της ΑΦΕΤ και του Διευρυμένου Προεδρείου, προκειμένου κάτι να αλλάξει στους κανονισμούς του σώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί το θέμα της κατάργησης των αν μη τι άλλο, είναι επιμερισμένη ευθύνη η δική μας και λίμπε. Η κατάργηση των θεωρήσεων αποτελεί εργαλείο εξωτερικής πολιτικής, άρα δεν πρέπει να το αναλάβει μια επιτροπή η οποία ασχολείται με τα εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα, τα τεχνικά, τα βιομετρικά ε, διαβατήρια και οι σχετικές συμφωνίες είναι θέματα δικά μας. Η δικιά μας η φωνή πρέπει να ακούγεται κατά πρώτον ή τέλος πάντων εξίσου με τη φωνή της Λίμπε. Και τώρα περνάω στην περίπτωση της Ουκρανίας. Εγώ δεν γνωρίζω καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα που είναι έτοιμη να πληρώσει με το αίμα της για να ακουστεί η ευρωπαϊκή της φωνή. Δεν ξέρω καμία ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα έκανε μεταρρυθμίσεις με τέτοια αποφασιστικότητα όπως κάνει η Ουκρανία να φτάσει σε πόλεμο, να τεθεί σε ομοιρία όπως έγινε στην περίπτωση της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Οπότε θα ήταν δίκαιο να επιτρέψουμε στους πολίτες, τους Ουκρανούς, να ταξιδεύουν χωρίς θεωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχρόνως θα ήταν και ένα ισχυρό μήνυμα και αναγνώριση των όσων έχουν λάβει χώρα στην Ουκρανία μετά τα γεγονότα της πλατείας Μαϊντάνου. Είναι μια διαδικασία επίσης για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης που έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι προχωράει. Για το λόγο αυτό λοιπόν και έχοντας την άποψη ότι έχει τηρήσει όλα τα κριτήρια του σχεδίου δράσης η Ουκρανία και ότι πολιτικά αξίζει τη συμβολική αυτή πράξη της αναγνώρισης πρέπει να αποδώσουμε το καθεστώς κατάργησης θεωρήσεων στην Ουκρανία χωρίς άλλη καθυστέρηση. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση ενώ και την υπόθεση της συμφωνίας με την Τουρκία. Η Ουκρανία έχει πετύχει πολλά. Και αυτό που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι παραμένει πιστή στις δημοκρατικές αξίες σε αντίθεση με αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς για μια άλλη χώρα όπως είναι η Γεωργία. Παρά λοιπόν την τήρηση των κριτηρίων και των προδιαγραφών και αξίζοντας την κατάργηση των θεωρήσεων, Συγχρόνως πρέπει να πούμε ότι οι διαδικασίες μεταρρύθμισης πρέπει να συνεχιστούν και να περάσουν σε πιο έντονο ρυθμό τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς κλπ. Γι' αυτό θα ήταν καλό να αναφερθούν οι προσπάθειες που κάνει η Ουκρανία στην έκθεση, αλλά να μιλάμε και για έναν μόνιμο μηχανισμό που θα διασφαλίζει ότι η διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Αυτός ο ειδικό μηχανισμός θα ήταν σαν την ε, σπάθα του Δαμοκλέους. Αλλά ή μάλλον ο μηχανισμός αναστολής είναι σαν σπάθα Δαμοκλέους, αλλά δεν είναι κάτι αποτελεσματικό, γιατί έχει να κάνει μόνο με τη μετανάστευση. Ενώ εδώ πέρα μιλάμε για γενικότερα κριτήρια. Οπότε θα χρειαζόταν κάποιο άλλο είδους μηχανισμός. Πάντως, ο προτινόμενος μηχανισμός ελέγχου που αποτελεί μέρος της πολιτικής μας γειτονία δεν πρέπει να αναβληθεί, αλλά θα πρέπει να συμπληρωθεί αργότερα. Η προσπάθεια της Ουκρανίας είναι χωρίς προηγούμενο. Οπότε, έλεγχος, ανταμοιβή, για τις μέχρι τώρα προσπάθειες, αλλά συγχρόνως και ενθάρρυνση. Όλα αυτά χρειάζονται για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην εισεγγελία, στο δικαστικό σώμα, στην ενίσχυση των θεσμών κράτους δικαίου. Γνωρίζουμε ότι οι προσπάθειες είναι τεράστιες, το αναγνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως οι αλλαγές και ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μένουν ακόμα πράγματα να γίνουν. Συνεπώς, η κατάργηση των θεωρήσεων πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για την Ουκρανία προκειμένου αυτή να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις της και να πετύχει τους πολιτικούς της στόχους. Επίσης, οι πολίτες της Ουκρανίας βλέπουν μια τέτοια χειρονομία σαν μια αναγνώριση του θάρρους που απέδειξαν. Η Ουκρανία δεν θα πρέπει να είναι θύμα εξαιτία συμφωνιών που κάνουμε με άλλε χώρε όπω την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό το θέμα τη θεω... της τη θεώρηση πρέπει να δοθεί για την Ουκρανία και να μην περιμένουμε να γίνει πρώτα για την Τουρκία και μετά για την Ουκρανία. Ευχαριστούμε κύριε Βόλσκι. Τώρα εκ μέρου του ΕΛΚ η κυρία Αντρακανιέτη έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω με όλους αυτούς που πιστεύουν ότι η κατάργηση της θεώρησης είναι ένα από τα κυριότερα κίνητρα για την κυβέρνηση της Ουκρανίας προκειμένου αυτή να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Αποτελεί και το στοιχείο κλειδί όσον αφορά τα κίνητρα αυτή τη στιγμή. Οι Ουκρανοί εξάλλου το αξίζουν και οι αρχές έχουν κάνει τα πάντα για να συμμορφωθούν με τις τεχνικές και νομικές προδιαγραφές και δεν αποτελούν και καμία τεράστια μεταναστευτική δυσκολία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου έχουν προχωρήσει σε πολλές σημαντικές και λογικές ε, μεταρρυθμίσεις με κοινή λογική. Θα λέγω ότι καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν σε θέση να εφαρμόσει τόσο αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις όπως έγινε από την Ουκρανική κυβέρνηση. Η καθυστέρηση στην απόδοση του καθεστώτος κατάργησης των θεωρήσεων από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία εσωτερικών θεμάτων των ευρωπαϊκών χωρών ήταν ένα χτύπημα για τι δυτικοευρωπαϊκέ ε, δυνάμει ε, τόσο στην Ουκρανία αλλά και σε όλες τις χώρες της ανατολικής μας εταιρική σχέση. Δεν πρέπει λοιπόν με τίποτα να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί το θέμα της κατάργησης θεωρήσεων για να πιέσει να τηρηθεί η συμφωνία των, του Μίνσκ από πλευρά των Ρώσων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σάντρα. Η κυρία Γκόμες έχει τώρα το λόγο, του των σοσιαλιστών παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέρφους που πήραν το λόγο πριν από μένα για το ότι η Ουκρανία πρέπει να αξιολογηθεί βάσει των δικών της επιτευγμάτων βάσει των όσων έχει κάνει για να τηρήσει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την κατάργηση των θεωρήσεων. Πήγα στην Ουκρανία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και συμμετείχα εκεί με τη Ρεμπέκα Χάρμς και την Σόφιν Χετφέλτ, τους συναδέρφους μας, σε Pride March. Και πρέπει να σας πω ότι πήγε πολύ καλά. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω πάει σε διαδήλωση με τόσο πολλούς αστυνομικούς που ήταν με το μέρος, θέλω να πω, των ε, ανθρώπων που έκαναν την πορεία, έτσι. Και αυτό από μόνο του αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα ότι οι αρχές της Ουκρανίας, τις βασικές ελευθερίες και τα βασικά δικαιώματα και τα, την ισότητα μεταξύ των πολιτών, τα παίρνουν πολύ σοβαρά και τα δικαιώματα των ε, ΛΟΑΔ. <coughs> Συμμορφώνονται δηλαδή όντως με τις ε, ευρωπαϊκές προϋποθέσεις. Πήγε πολύ καλά λοιπόν αυτή η πορεία ε, των ΛΟΑΔ. Τώρα, συζητήσαμε και φυσικά και υπάρχουν τομείς όπου ακόμα μπορούν να βελτιωθούν. Ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως των φυλακισμένων στο Τόμπας και δεν μιλάω για αυτούς που κρατούνται από δυνάμεις οι οποίες δεν ελέγχονται από τους Ρώσους, γιατί προφανώς τότε δεν ελέγχουν η Ουκρανική κατάσταση. Μιλάω για τους κρατούμενους από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Όμως, πράγματι, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι τεράστια αν τις συγκρίνουμε με την κατάσταση την εποχή της πλατείας Μαϊντάν. Όντως, πρέπει να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις. Θα ήταν κρίμα να μην γίνει αυτό. Και θα ήταν κρίμα για τις ευρωπαϊκές αξίες αν δεν ανταμείβαμε την Ουκρανία για τόσα έχει πετύχει μέχρι τώρα. Η περίπτωση τώρα της Τουρκίας δεν αποτελεί λόγο να καθυστερήσουμε. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι λόγος να επιταχύνουμε ε, τα πράγματα με την Ουκρανία για να δείξουμε ότι ανταμείβουμε πράγματι αυτούς που βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Και ότι δεν ε, κλείνουμε τα μάτια στα τεράστια ε, προβλήματα και τις οπισθοχωρήσεις που έχουν γίνει στην Τουρκία όσον αφορά το σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεχάγης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τεμεσμάκερ έχει τώρα, εκ μέρους του ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να πω ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, ε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω τέτοια, γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Η ομάδα μας, το ECR, στηρίζει απόλυτα το καθεστώς κατάργησης των θεωρήσεων για την Ουκρανία. Το σχέδιο δράσης προτάθηκε το 2010 Είμαστε τώρα έξι χρόνια αργότερα και μία επανάσταση αργότερα. Μετά το Μαϊντάν έγιναν γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία. Η επανάσταση αυτή των αξιών και οι δημοκρατικές εκλογές έδειξαν ότι ο λαός της Ουκρανίας έχει επιλέξει ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τον εαυτό του. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέλει πραγματικά η συμφωνία σύνδεσης ε, και ελεύθερο συναλλαγών και θέλει να πετύχει, τότε πρέπει να καταργηθεί η βίζα, οι θεωρήσεις για τους Ουκρανούς πολίτες που έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Η Ουκρανία έχει επιλέξει την Ευρώπη και ελεύθερα αποφασίζει που θέλει να πάει και θέλει να αντιμετωπίσει τον ε, άγριο γείτονά της εξανατολών. Το πλαίσιο λοιπόν είναι τέτοιο που πρέπει να προχωρήσουμε και δεν πρέπει να το συνδέσουμε με άλλες χώρες και με άλλες περιπτώσεις. Η κάθε χώρα και ο κάθε φάκελος χώρας πρέπει να κριθεί βάσει των συγκεκριμένων επιτευμάτων και όχι σε σχέση με άλλες χώρες. Συνεπώς, να ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιτέλους πρέπει να δείξουμε στους Ουκρανούς τι δικαιούνται. Χρειάζεται βέβαια καταπολέμηση της διαφθοράς, ε, σεβασμός του κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία παραμένουν στο τραπέζι. Υπάρχουν δυσκολίες και για την πλήρη τήρηση των ε, κριτηριών. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μάρκ. Η Πέτρα Αστροβίτσιος τώρα, εκ μέρους της Άλντε. Παρακαλώ, ο κύριος Αστροβίτσιος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σήμερα συζητούμε θέμα το οποίο είναι ενδεικτικό με τον καλύτερο τρόπο για το τι γίνεται με τις συμφωνίες σύνδεσης οι οποίες προκειμένου απέδωσαν ήταν κίνητρο για μεταρρυθμίσεις για αλλαγή και για διαφορετικούς μετασχηματισμούς Επομένω έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι. Είδαμε σε μία διετία τι έγινε υπό συνθήκε πολύ δύσκολε. Οπότε και τονίζω για άλλη μια φορά συμφωνώντα με τους προελίσσαντες. Η Ουκρανία αξίζει την αναγνώριση. Και με το παραπάνω γιατί αυτέ οι μεταρρυθμίσει συνετελέστησαν υπό συνθήκε πολέμου, επιθετικότητας, κατάληψης της επικρατείας του και δύσκολη οικονομική κατάσταση παρόλα αυτά. Επομένω, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να υπάρχει η ισχυρή θέληση για αλλαγή, για μεταρρυθμίσεις, οπότε όλα αυτά τα οποία ε, αξίζουν να προχωρήσουμε στην υπόθεση της απελευθέρωσης της θεωρήσης διαβατηρίου και είδαμε διάφορες τομιακές ε, μεταρρυθμίσεις. Να το αναγνωρίσουμε και να τα αναγνωρίσουμε ένα προς ένα όσα επιτεύχθησαν και εγώ πιστεύω επομένω ότι δεν θα πρέπει να ομαδοποιούμε τη θεώρηση των πραγμάτων. Άρα θα πρέπει περιπτωσιολογικά να αντιμετωπίζουμε τα επιτεύγματα. Θα πρέπει να συμφωνήσετε συναδελφοί ότι ο μηχανισμός αναστολής που υπέστη την τροποποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου ήταν κάτι το αναπόφευκτο υπό τις παρούσες συνθήκες. Όχι, γιατί αυτό είναι νερό στον μήλο αυτών που δεν θέλουν απελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου. Θα πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο αυτών που μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή χωρίς χωρί του διαβατηρίου. Αυτό είναι απόφευκτο, αλλά ο μηχανισμός αναστολής είναι κάτι το οποίο πρόκειται να ρυθμίσει τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της θεώρησης διαβατηρίου. Εκεί θα λειτουργήσει ο μηχανισμός αναστολής. Οι χώρες οι οποίες ε, έχουν περάσει από αυτές τις συμφωνίες ε, και που συμμορφούνται προς αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόβλημα. Επομένως, οι ουκρανικές μεταρρυθμίσεις, ιδίω όσον αφορά την αστυνομία, όσον αφορά την δικαιοσύνη, ε, που μέχρι και πολύ πρόσφατα συνετελέστησαν, Νομίζω ότι δίνουν και ουστά στην συμφωνία, οπότε και εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε την εμπιστοσύνη μας. Την χρειάζεται τη βοήθειά μας η χώρα για το άμεσο μέλλον, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Άρα θα πρέπει να τίνουμε χείρα αλληλεγγύης προς τη χώρα τώρα. Σε ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Πλέγκοβης, για τα όσα μας είπες και τώρα ο κύριος Κόρβιν Μίκη έχει το λόγο. Φυσικά. Οποιοςδήποτε φιλελεύθερος θα υποστηρίξει τη φιλελευθερωποίηση και εγώ το ίδιο. Θέλω να στρέψω την προσοχή σας σε δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να υπάρχουν ελευθερία προξενικών θεωρήσεων για όλους τους Ουκρανούς, ώστε το μισό της Ουκρανίας που πρόσχεται στη Ρωσία να μπορεί να πάει στη Δύση και οι Ουκρανικές μαφίες και οι μυστικές υπηρεσίες πολλές φορές ταυτίζονται οι δύο αυτοί ευαγείς φορεί είναι πολύ καλή στο να παραποιούν ε, διαβατήρια, ταυτότητες κτλ. Αν υπάρξει λοιπόν πλήρης φιλελευθερωποίηση, <coughs> σε δύο χρόνια δεν θα έχουμε 40 μοναχα Ουκρανούς, αλλά 50-60 εκατομμύρια Ουκρανούς που θα έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε πάντα δημιουργικός σε αυτά τα θέματα, πιστεύω. Ο κύριος Στέτινα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χθες συζητήσαμε το θέμα των προξενικών θεωρήσεων για την Γεωργία. Σήμερα, σήμερα το συζητούμε για την Ουκρανία. Να επιστήσω όμως την προσοχή σας σε μια μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών της Γεωργίας και της Ουκρανίας η Γεωργία έχει ένα ε, στρατό κατοχής της επαρχίας της Αυχαζίας και της Σωσετίας. Έχουμε δύο παγωμένες σειράξεις εκεί. Ενώ η Ουκρανία είναι σε μια θερμή πολεμική σύραξη με 10.000 νεκρούς. Έχουμε 1,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους στην Ουκρανία. Το το Τίρασπολ και το Ντόνμπας είναι περιοχές όπου πεθαίνουν οι νέοι και σκοτώνονται κάθε μέρα. Πολλοί χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη μεταξύ άλλων. Το Μάιο μαζί με τον κύριο Σφάτσεμπερ, ο οποίος ήταν ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας, πήγαμε στο Ντόνμπας και συναντήσαμε τον κύριο Σαμπρέτσκι ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει λόγω της ε, εισβολής των Ρώσων. Και το γεγονός ότι μόνο δύο Ευρωπαίοι πολιτικοί ήταν παρόντες εκεί στο Τον ενθαρρύνει πάρα πολύ το λαό της περιοχής, ο οποίος είναι ζητάει πάντα την ε, υποστήριξη των ε, Ευρωπαίων. Το να δώσουμε λοιπόν ένα καθεστώς προξενικής, ε, μάλλον εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί προξενικέ θεώρησει είναι κάτι πολύ θετικό για αυτού οι οποίοι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και αγωνίζονται για την ελευθερία του. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πίτσουλα έχει το λόγο. Είναι φυσικά σκιώδη συζητή για του σοσιαλιστέ, αλλά δεν μου το είχαν υποδείξει αυτό. Ο Τονίνο λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η διαδικασία φιλελευθερωποίησης για τι προξενικέ θεωρίε έχει ξεκινήσει σε συνθήκε πολύ διαφορετικέ από ό,τι προβλεπόταν πριν από 8 χρόνια. 22 Νοεμβρίου του 2010 η Κομισιόν παρουσίασε ένα σχέδιο δράση σε σχέση με την φιλελευθερωποίηση στα θέματα αυτά. Υπήρξε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είχαν καθοριστεί και είχαν οργανωθεί σε τέσσερις ομάδες με στόχο να επιτευχθεί η εναρμόνιση σε νομοθετικό πλαίσιο και να εξασφαλιστεί η μόνιμη εφαρμογή των μέτρων αυτών. Έγινε η έγκριση της κατάλληλης νομοθεσίας, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί με πιστικό τρόπο. Πέραν όμως αυτών των κριτηρίων και της ε, καταληκτικής ημερομηνία, χρειαζόμαστε να έχουμε το σωστό πνεύμα για τους πολίτες Ουκρανίας που πλήττονται από την εξωτερική ε, επιβολή και τις εσωτερικές ανταρσίες. Η φιλελευθερωποίηση λοιπόν του καθεστώτος υποξενικών θεωρήσεων θα μας δώσει και πάλι την ευκαιρία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξη προ το λαό της Ουκρανίας. Και γι' αυτό εγώ προσυπογράφω απόλυτα την άποψη του εισηγητή ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την εξαίρεση όσο το δυνατόν ευρύτερη για τους πολίτες της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι ε, παραγνώριση της άποψης πολλών από τους συμπολίτε μας, όπως είναι οι κατοχωρίτες οι Ολλανδοί. Γιατί πάντα μπορεί να αρθεί ένα ε, καθεστώς ελευθερίας από προξενικές θεωρίες. Περνάμε μια φάση κόπωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή η κόπωση δεν πρέπει να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό στην προσπάθειά του να μπορέσει να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε άλλου ομιλητέ, αλλά έχουμε τον κύριο Κούκαν, ο οποίο θέλει και αυτό να λάβει το λόγο. Μία πρόταση μονάχα θέλω να πω, για να προσθέσω και τη δική μου φωνή σε αυτού οι οποίοι υποστήριξαν την ιδέα του εισηγητή, του κύριου Βόλσκι. Νομίζω ότι η συζήτηση ε, κατέδειξε ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για την κατεύθυνση του εισηγητή και η μόνη έκκληση που θέλω να κάνω σε όλους είναι ότι τώρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να γίνει πραγματικότητα αυτή η απελευθέρωση των προξενικών θεωρήσεων χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Κάποιο άλλο θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Δίνω και πάλι το λόγο στον εαυτό μου, αλλά σε διαφορετική ιδιότητα, ω Προέδρο τη Αντιπροσωπείας με την Ουκρανία, για να τονίσω ορισμένα σημεία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι το θέμα της φιλελευθερωποίηση για τις βίζες σε ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπιστεί από στρατηγική έποψη. Κάθε δύο μήνες ουσιαστικά πηγαίνω στην Ουκρανία και θα έχω και πάλι επαφές με Ουκρανούς ε, εμπειρογνώμονε, κοινοβουλευτικού, φοιτητές ε, κτλ. το Σαββατοκύριακο αυτό. Μπορώ να σας πω ότι διαβλέπω αυτή την ματέωση, την απογοήτευση που νιώθουν επειδή καθυστερούμε. Δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε δι, ούτε αξιόπιστο το να καθυστερούμε. Ανεξάρτητα από τις αμφιβολίες μας, ήδη αντιλαμβάνεται η καθυστέρησή μας ως κάτι αρνητικό για την ευρωπαϊκή διαδικασία μια χώρας η οποία ευρέθη κάτω από ε, επίθεση και εισβολή. Έχουμε μια ηθική υποχρέωση προς την Ουκρανία. Πρέπει να σας πω επίσης ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είτε είμαστε οι βουλευτέ τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, είτε τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είτε από την Επιτροπή Πολιτισμού, αποτελούμε ένα θεσμικό όργανο και πρέπει να δράσουμε ενωμένοι. Μια παρόμοια συζήτηση αυτή τη στιγμή γίνεται στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στο Συμβούλιο ε, Δημοσίων Ελευθεριών, Εσωτερικών και Δικαιοσύνη. Σήμερα θα συζητήσει το Συμβούλιο και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί θα έχει σαφείς επιρροές στη δυναμική των σχέσεων μας με την Ουκρανία. Η <clears throat> διαδικασία αναστολής που προβλέπεται φυσικά επηρεάζει πολύ τις θέσεις των χωρών αυτών. Γι' αυτό έχουμε πέντε από τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου της ε, Ουκρανίας που έρχονται σε μια συζήτηση με την Επιτροπή μας. Σας παρακαλώ λοιπόν όσοι θέλουν και ενδιαφέρονται να είναι εδώ για να ακούσετε ποια είναι η δική τους αντίληψη, ο διεκτόπος που βλέπουν αυτή τα πράγματα και γιατί πιστεύουν ότι ο Επίτροπος ε, Χάν και η Κομισιόν ε, τόνισαν ότι είχαν εκπληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα. Δεν το σκέφτηκαν μοναχά και να το πούνε αμέσως μετά από μια μέρα. Μετά από μια ενδελεχή ανάλυση των ερεσιμοτήτων και των κριτηρίων μονάχα στο φάκελο της φιλελευθερωποίησης των ε, προξενικών θεωρήσεων, μόνο τότε το έκαναν και είπαν ότι έχουν εκπληρωθεί όλα αυτά. Κάτι ακόμα που δεν αναφέρθηκε από πολλούς. Έχουμε 1,5 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους στην <clears throat> Ουκρανία. 1,5. Είναι περισσότερο, περισσότερο αυτό το νούμερο από όλους αυτούς που είδαμε να έρχονται από τη Μεσόγειο ως πρόσφυγες στην Ευρώπη πέρσι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να το παραμελήσουμε. Η Ουκρανία έχει δείξει την ικανότητα να απορροφήσει μέσω στους θεσμικούς τρόπους και με την αλληλεγγύη μεταξύ των απλών ανθρώπων όλους αυτούς οι οποίοι χρειάστηκε να φύγουν από τις προσωρινά ε, περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, του Ντονέσκ και άλλων περιοχών. Είναι λοιπόν δική μας <clears throat> θεσμική και πολιτική ευθύνη να πράξουμε τα απαραίτητα. Θα πρέπει να δείξουμε στους συναδέλφους μας στην Ουκρανία μέσω των πολιτικών ομάδων και εδώ βασίζομαι στην θέση όλων των σκιωδών συγητών που μπορούν να πείσουν τους ομολόγους τους στις πολιτικές τους ομάδες πρέπει να δείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ενότητα για το θέμα αυτό. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τι διαδηλώσει του Μαϊντάν. Είναι μεγάλε οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί στην Ουκρανία. Η Συμφωνία <clears throat> Σύνδεσης αντιμετώπισε μια μικρή καθυστέρηση και λόγω της, ε, του δημοψηφίσματος ε, των κάτω χωρών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τονίσουμε τη σημασία την πολιτική που έχει το καθεστώ ελευθερίας από προξενικέ θεωρίες. Ας αρθούμε στο ύψος των πολιτικών προσδοκιών ως κοινοβούλιο και ως εκλεγμένη κοινοβουλευτική. Υποστηρίζω λοιπόν απόλυτα αυτά τα οποία είπε ο εισηγητής και πιστεύω ότι και οι συναδελφοί μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα δείξουν και αυτή την απαραίτητη σπουδή ώστε να περατωθεί αυτή η έκθεση και να έρθει στην ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τη δική μας επιρροή για να δώσουμε το μήνυμα αυτό υπευθυνότητος και στα κρατημέλη, στο Συμβούλιο πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ε, απόφαση. Μπορώ έτσι να κλείσω το θέμα αυτό τη σημερινή διάταξη, εκτό αν ο Γιάτσεκ θέλει να πει κάτι που προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Σύμφωνο απόλυτα με τα συμπεράσματά σας, υπό τη διπλή σας ιδιότητα και ως πρόεδρος δηλαδή, και ως πρόεδρος της αντιπροσωπής για τις σχέσεις μας με την Ουκρανία. Το μόνο που θα είχα να προσθέσω είναι ότι ελπίζω πως ε, ομόφωνα θα ζητήσουμε την απόδοση του καθεστώτος ε, κατάργησης θεωρήσεων στην Ουκρανία. Το θέμα δεν είναι μόνο δηλαδή να επηρεάσουμε του συναδέρφους μας στις διάφορες επιτροπές, είναι και θέμα κυβερνήσεων. Έχουμε την ευθύνη να πούμε στις ε, κυβερνήσεις μας, είτε είμαστε στην αντιπολίτευση είτε όχι, ποια είναι η θέση μας εδώ. Γιατί θα ήταν μοιραίο, θα ήταν πολύ κακό εξαιτία ε, της πολυπλοκότητας της τουρκικής συμφωνίας, για να το πω έτσι ίδια να χρησιμοποιηθούν επιχειρήματα κατά της Γεωργίας ή της Ουκρανίας. Θα χαθεί η υπόθεση της ε, Ουκρανίας θα αναβληθεί και καταλαβαίνετε πόσο αρνητικό θα είναι, όπως ακριβώς το περιγράψατε. Οπότε να κάνουμε αυτό που προτείνατε και συγχρόνως να ζητήσουμε από τους επικεφαλείς των ομάδων μας και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου μας να εκφραστούν έντονα για να προσθέσουν και αυτή τη φωνή τους στα αποτελέσματα του Συμβουλίου. Να μην είναι μόνο δηλαδή από το επίπεδο της Επιτροπής μας ή των Επιτροπών γενικά, αλλά να έρθει η φωνή ερθει φωνη αυτη και από πιο ισχυρές θέσεις. Και στις χώρες μέλη βέβαια να επηρεάσουν όπως μπορούν οι ευρωβουλευτές τα πράγματα, ώστε να επηρεαστεί η κατάσταση και να καταλάβει και η κοινή γνώμη ότι πολιτικά δημιουργούνται δυσκολίες και κοστίζει αν ε, δεν προχωρήσει η συμφωνία αυτή για την κατάργηση των για τους Ουκρανούς. Να ενισχύσουμε το μήνυμά μας όσο μπορούμε δηλαδή. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαριούς Φόλσκι. Ο πρόεδρος Σούλτς έχει ήδη λάβει επιστολή από τον πρόεδρο Ρουνταράντα όσον αφορά το επίγον της απόφασης. Η Επιτροπή. Α, συγγνώμη, δεν είχα αντιληφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε το λόγο. Παρακαλώ, για πείτε μας από ποια γενική διάθεση. Είμαι Καρμέλα Σμίτ από την DG Home. Είμαι αρμόδια για την πρόταση αυτή όσον αφορά την κατάργηση θεωρήσεων με την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας στην πρότασή μας. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι η ομάδα εργασίας για τις θεωρήσεις, που σε 30 λεπτά θα αρχίσει να συνεδριάζει, θα συζητήσει τις διάφορες προτάσεις μία-μία όσον αφορά την κατάργηση θεωρήσεων. Δεν πάνε δηλαδή πακέτο για όλες τις χώρες, για κάθε μία χωριστά. Σημείωσα ότι ζητούν οι ευρωβουλευτές την εισαγωγή ενός μηχανισμού ελέγχου της ε, συνέχειας των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για την τήρηση του κράτους δικαίου, ακόμα και όταν έχει αποδοθεί η διευκόλυνση αυτή κατάργηση ιστορίσεων για τους Ουκρανούς. Έχουμε λοιπόν και την πρόταση για τον μηχανισμό αναστολής θα υποβληθεί η πρόταση αυτή στη ΛΥΜΠΕ από τον κύριο Ντίες Ντεμέρα, τον εισηγητή. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι η απόφαση για την κατάργηση θεωρήσεων ε, στους Ουκρανούς δεν πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να εγκαθιδρυθεί ένας τέτοιος μηχανισμός. Πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσουμε, δεδομένου ότι όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσης για την Ουκρανία προκειμένου να καταργηθούν οι θεωρήσεις για τους Ουκρανούς έχουν ε, υλοποιηθεί. Πρόεδρο, συγγνώμη, βλέπετε, εγώ κοίταζα προς την άλλη μεριά και δεν ε, αντιλήφθηκα ότι οι Γενικές Διευθύνσεις Home και Near ε, βρίσκονται σε 20 μέτρα απόσταση. Ευχαριστώ πάντως για τόσα μας είπατε για την ενημέρωσή σας. Σίγουρα θα βοηθήσει τις αποφάσεις μας. Τώρα υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στη γνωμοδότηση αυτή είναι 21η Ιουνίου. Όσοι λοιπόν θέλετε να υποβάλλετε προτάσεις μέχρι τότε. Καλώς και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αυτό είναι τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Εδώ είναι ήτρε η αρμόδια επί της ουσίας με αεριο εδω ειναι ητρε η αρμοδια επι της επιτροπης η δικιά μας γνωμοδότηση είναι στα χέρια του κύριου Σάρις Βόλσκι, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα θέματα ενέργειας και στόλ. Έχετε το υλικό, την αιτιολόγηση και τη σημασία που έχει η κατοχήρωση της ασφάλειας εφοδιασμού αερίου. Οι διαφορετικές πηγές ο εφοδιασμός από διαφορετικές χώρες είναι ουσιώδες. Τα τελευταία χρόνια περάσαμε από κρίσεις που πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο κύριος Άριος Βόλσκι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακριβώ όπω και για την προηγούμενη εκθέση, επιτρέψτε να ξεκινήσω μια γενική παρατήρηση. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι αρμοδιότητα που ξεκίνησε το 2007 ε, ως αρμοδιότητα της ΑΦΕΔ γιατί το Κοινοβούλιο παρατηρήσε ότι υπάρχει ε, θέμα ενεργείας ασφάλειας όταν είχαμε το 6 και το 7 το, το, κόψιμο της παροχής ε, αερίου από τη Ρωσία προς την Ουκρανία και είπαμε ότι υπάρχει τέτοιο θέμα ασφάλεια. ασφάλειας και άρα θα πρέπει στα πλαίσια των έχουμε και να λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει το γραφείο της Επιτροπής μας ε, να ζητήσει να είναι κοινή αρμοδιότητα η τρεκή ΑΦΕΤ. Να μην έχουμε εμείς ε, συντρέχουσα απλώς ε, γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Και τώρα επί της ουσίας για δεύτερη φορά. Κάντε ησυχία συνάδελφοι παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ λίγα για δεύτερη φορά επομένω ασχολούμεθα με έναν κανονισμό που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια για πρώτη φορά. το στήσαμε πριν από 5 ή 6 χρόνια. Και υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα κείμενο το οποίο απήχε πολύ από το να είναι άρτιο οπότε και βελτιώσαμε σημαντικά το κείμενο αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο το τροποποιήσαμε, το αλλάξαμε και το βελτιώσαμε σημαντικά Ακριβώς πρόκειται για τον κανονισμό που πρόκειται τώρα να καταργηθεί με την τρέχουσα πρόταση. Πέρασαν 5 χρόνια και μπράβο που τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσθέσει ένα πολύ καλύτερο κείμενο. Οπότε και σήμερα ο ρόλος μας δεν είναι το να αλλάξουμε εκ βάθρων αυτό το κείμενο ή να, να, να Απλώς να επιφέρουμε κάποιες μικρές βελτιώσεις και βεβαίως ε, θα υπεραμεινθούμε της πρότασης της Επιτροπής σε σχέση με αυτούς που θέλουν να την ε, απονευρώσουν διότι αυτή η πρόταση όπως ήδη γνωρίζουμε ε, βρίσκεται ε, στο στόχαστρο κάποιων κύκλων. Επομένως, αυτός ο οργανισμός είναι κάτι το θετικό και εστιάζει σωστά στην πληροφορική συνεργασία και σε μηχανισμούς ασφαλείας και ο στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλαμβάνεται περισσότερο των ενεργειακών που συνδυάζονται και με τις εξωτερικές μας σχέσεις. Η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διακοπής ε, παροχής και να προστατευτεί ο καταναλωτής. Άρα θα πρέπει να φέρουμε κάποιες βελτιώσεις σε αυτά τα σημεία, να έχουμε προληπτική δράση, αλλά επίσης και ε, κάλυψη των ε, κατεπηγουσών περιπτώσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν σε σχέση με την υλοποίηση της ε, ρήτρας ελληνικής. Θα πρέπει να υπάρχει επίσης υλοποίηση ε, της ε, ρήτρας ε, για τα κατεπήγοντα και ακόμα μόνος δεν είναι τόσο στεγανό θα έπρεπε, το κείμενο. Άρα υπάρχει το θέμα ε, των ομαδοποιημένων προμηθειών και αυτό το έχει προτείνει επίσης το Συμβούλιο. Θα πρέπει να καλυφθούν όλες ένωσης με, από τους μηχανισμούς που προβλέπει το άρθρο 15 αυτό το οποίο εμεί θεωρούμε μεγαλύτερο πρόβλημα και το επισημαίνουμε έχει να κάνει με την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις συμβάσεις μεταξύ των εταιριών. Φανταστείτε, μια κατάσταση όπως σήμερα. Ο κύριος Πούτιν συναντά τον κύριο Γιούνκερ. Ο κύριος Πούτιν έχει στα χέρια του συμβάσεις για την προμήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το αφεντικό της Γκάσπρομ και όλα τα έχει υπόψη. του Στην άλλη μεριά του τραπεζιού, ο κ. Γιούγκερ που δεν έχει καμία σύμβαση. Εμεί τι θέλουμε. Θέλουμε κάποιον που μα εκπροσωπεί ω Ένωση να βρίσκεται σε τόσο αδύνατη διαπραγματευτική θέση έναντι τη άλλη πλευρά, η οποία όπω όλοι γνωρίζουμε καλά χρησιμοποιεί την ενέργεια, χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ω μέσο άσκηση εξωτερική πολιτική. Ε, αυτό θα πρέπει να αλλάξει επομένω σας καλώ να αναβαθμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενημέρωση που χρειάζεται ε, όσον αφορά το φυσικό αέριο, τις συμβάσεις με ε, τις ε, άλλες εταιρείε και βεβαίως την Gazprom. Προτείνεται επομένω ένας μηχανισμός εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε και δεν συμφωνώ ότι όλες οι συμβάσεις που είναι πάνω του 40% της ζωής να ε, αποκαλύπτονται. Όμως δεν είναι λογικό ενώ εμείς μιλούμε και ενεργούμε ε, να υπάρχει πανευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου να έχουμε ένα νομοθέτημα που αφορά μόνο την αγορά μιας χώρας. Αυτό είναι παράλογο, αυτό είναι τελείως ασύμβατο με τη λογική της ενιαίας αγοράς που θέλουμε. Επίσης, αυτή ε, η κατάργηση της διαβάθμισης τέλο πάντων ε, όταν έχουμε κάποιες χώρες που, για τις συμβάσεις που υπάρχουν για το πάνω το 40% των εισαγωγών ή της κατανάλωσης τότε έχετε πάρα πολλές χώρες βαλτικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία κλπ. θα αποκαλύψουν τις συμβάσεις, αλλά η Γερμανία, η Φιλανδία δεν θα αποκαλύψουν διότι έχουν ε, πάρα πολύ σημαντικές συμβάσεις, αλλά είναι κάτω του 40% της κατανάλωσης. Οπότε γι' αυτό αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε είναι αντίθετο στην ιδέα της ενιαίας αγοράς φυσικού αερίου. Είναι κάτι το άδικο, επομένως θα πρέπει να αντικατασταθεί ε, αυτό το 40% της, και θα πρέπει να υπάρχει αντί για το ποσοστό ένα νούμερο. Αυτό πάει να πει ε, κοινοτικό κεκτημένο. Ανταγωνισμός. Η πρακτική που ισχύει σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει κάθε συγχώνευση, κάθε εξαγορά πάνω από μια συγκεκριμένη αξία, σε νούμερο, σε έναν αριθμό. Δεν είναι σχετικός ο προσδιορισμός, ένα ποσοστό τέλο πάντων, της εθνικής αγοράς. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους σας προτείνω να βάλουμε 80 δις και 8, 8, 8 δις κυβικά μέτρα. 8 δις κυβικά μέτρα. Οπότε, όποτε υπάρχει υπέρβαση, να υπάρχει σχετική ενημέρωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το 40% να είναι απλώς επικουρικό για κάποιες χώρες που είναι ενεργειακές νησίδες όπως οι βαλτικές χώρες. Για αυτό αυτή είναι η βασική μας ε, διαφορά. Θέλουμε αυτό να αλλάξει. Είναι αυτό που ορίζεται στο άρθρο 13. Επομένως, συνοψίζω. Κατά τη γνώμη μας και σύμφωνα με τις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει, θέλουμε να αναβαθμιστεί και να υπάρξει περιφερειακή προσέγγιση. Γιατί τώρα, όπω ξέρετε, πολλέ μεγάλε χώρε αμφισβητούν μια τέτοια προσέγγιση και πίσω από αυτέ τι χώρε κρύβονται ισχυρέ εταιρείε θα πρέπει να εναρμονίσουμε την προστασία του καταναλωτή και να μην είναι πιο σημαντικές οι εθνικές ρυθμίσεις από την περιφερειακή διάσταση. Να μην υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος θα παραλύσει την περιφερειακή συνεργασία και την υλοποίηση του οργανισμού. Επομένως, θα πρέπει το Συμβούλιο να δώσει εντολή στο, στην Επιτροπή, ούτως ώστε αν δεν ε, ε, υπάρξει συμφωνία με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να είναι δυνατόν Εάν δεν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους, να ενεργοποιείται η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών. Και γι' αυτό Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο φιλόδοξη σε αυτό το μέτωπο σε σχέση με κάποια κρατημέλη που δεν θέλουν αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Θέλουμε περισσότερη ενεργειακή διπλωματία και σας παραπέμπω στην έκθεση της ΑΦΕΤ που ε, ε, ολοκληρώθηκε το 2007 όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Επίσης, τέλος, θέλουμε να έχει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους ε, ενουσιακού παρόχους, ε, τις ε, ενουσιακές εταιρείες και να μην είναι σκλάβοι των μονοπωλίων οι καταναλωτές και λοιποί χρήστες φυσικού αερίου πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Σάρις Ο κύριος ε, Πίτσουλα, ο οποίος είναι σχεδόν συγητής, τώρα θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το νόημα αυτής της νομοθετικής πρότασης είναι να δώσουμε μια εγγύηση ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις διακοπές τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο ή την έκτακτη ζήτηση αν όλοι εξαρτώνται από μία πηγή μονάχα τροφοδοσίας, υπάρχει πάντα η δυνατότητα της διακοπής της τροφοδοσίας. Ο κίνδυνος αυτός μιας διακοπής της τροφοδοσίας δεν αφορά μονάχα ένα κράτος μέλος, αλλά πολλά κράτη-μέλη παράλληλα. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτήν την πρόταση για τη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας που να βασίζεται σε ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα οι καθαρά εθνικές αξιολογήσεις των κινδύνων δεν είναι πια τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Η βασική αρχή λοιπόν θα πρέπει να είναι η αρχή της αλληλεγγύης, βάσει της οποίας σε τελική ανάλυση οι γείτονε χώρες σε περίπτωση μιας κρίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν την απαραίτητη τροφοδοσία με φυσικό αέριο των οικοκυριών ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό κείμενο. Είναι μια πραγματικά ευρωπαϊκή θέση και την υποστηρίζω απόλυτα. Θα, ήθελα να πιστέψω ότι αυτή η πρόταση μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αν έχουμε σαφέστερους ορισμούς και πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ε, λειτουργία του μηχανισμού αλληλεγγύης και καλύτερο συντονισμό. Είναι χρήσιμο επίσης να αναφερθούμε και στις προθεσμίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ε, ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού και να εξασφαλίσουμε την πλήρη συνεργασία των εμπλεκομένων κρατών μελών. Και είναι θετικό να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την περιφερειακή συνεργασία με αυτόν τον τρόπο και να συμπεριλάβουμε και όμορες χώρες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και σαφείς υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην Ένωση Ενέργειας. Ο Μάρκ Ντέμεσμέκερ τώρα για, τους, για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στην αλλαγή που θέλουμε για την ενέργεια, προκειμένου να πάμε σε πράσινη ενέργεια, σίγουρα για ένα χρόνο το αέριο συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο. Μπορεί να είναι ορυκτό, αλλά τέλο πάντων δεν είναι τόσο επιβλαβές ε, όσο άλλα ορυκτά. Φυσικά όλα αυτά προκειμένου να φτάσουμε στις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Πολλές φορές χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο και σε εταιρείε και στα σπίτια για να ζεσταθούμε. Και όλοι ξέρουμε ότι οι προβλέψεις ε, για την προμήθεια των εφοδιασμό φυσικού αερίου μερικές φορές μας έχει οδηγήσει σε πολιτικά παιχνίδια. Ε, τα είδαμε και με την Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Οπότε η Επιτροπή μας Εξωτερικών Υποθέσεων είναι η κατάλληλη για να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Τώρα πώς αντιστέκεται σε γεωπολιτικές εξωτερικές πιέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται συντονισμό μεταξύ μας, συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή από αυτού. Όντω, η Ενεργειακή Ένωση είναι ένα μέσο για να έχουμε περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μέτρα όσον αφορά τον εφοδιασμό, έτσι όπω τα έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα υπάρχουν τώρα διάφορα ζητήματα που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην γνωμοδότηση. Θα περιοριστώ σε τρία. Πρώτον, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι κανόνες ανταγωνισμού γίνονται σεβαστοί. Πρέπει αυτό οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα περιθώριο για παιχνίδια από δεσπόζουσα θέση στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε συνομιλίε με την Ουκρανία, με την Gazprom να οδηγήσουν ώστε ο εφοδιασμός στην Ουκρανία ρωσικού φυσικού αερίου να μην αποτελεί ένα μέσο εκβιασμού. Και τρίτον, αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη αποτελεί το κέντρο αλλά και τη δύναμη της Ενεργειακής μας Ένωσης. Πρέπει να στηρίξει η Επιτροπή μόνο προγράμματα τα οποία συνάδουν απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θα υποβάλω τροπολογίες όσον αφορά τα τρία αυτά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mark. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αουστρεβίτσιος. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα βασικό στοιχείο της γενικής ασφάλειας. Το θέμα αυτό όμως ε, δεν αντιμετωπίζει αρκετά από τους πολιτικούς, ενώ οι εμπλεκόμενοι στον χώρο της ενέργειας πάντα προσπαθούν να το επιτύχουν. Έχουμε δει κάποια ενθαρρυντικά βήματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την αναγνώριση ενεργειακής ασφάλειας ως σημαντικής πτυχής της γενικής έννοιας της ασφάλειας. Εγώ θα έλεγα ότι έχει υπάρξει μια αφύπνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Αν διαβάσετε το σχέδιο γνωμοδότηση που παρουσιάστηκε από την Κομισιόν, θα δείτε πολλά τεχνικά σημεία βέβαια και όπως ε, είπε ο κύριος Σάρις Φόλσκι, φαίνεται υπερβολικά πολύπλοκο με υπολογισμούς, με περιγραφές κτλ. Πίσω όμως από αυτές τις τεχνικές παρουσιάσεις υπάρχουν σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχίζουν όπως το παρελθόν για τα ενεργειακά θέματα, όταν μεγάλες εταιρείες και μεγάλες χώρες παρουσιάζανε το θέμα της ενέργειας σαν κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική πολιτική, αλλά μόνο με το επιχείρημα. Όχι. Έχουν οριμάσει λοιπόν οι συνδίκες για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε αυτή την προσέγγιση και να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς μια πιο συνεκτική ευρωπαϊκή ενεργειακή ένωση και πολιτική. Θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγέ και από τι δύο πλευρέ, και από την πλευρά τη ζήτηση και από την πλευρά τη προσφορά. Μεγαλύτερη συνεκτικότητα για την προσφορά και καλύτερη συνένωση τη ζήτηση. Εάν το πετύχουμε όλο αυτό, θα έχουμε πραγματικά μια ενεργειακή ένωση. Λέγοντα αυτό όμω, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο σε ό,τι αφορά την πρακτική εφαρμογή όλων αυτών των προνοιών. Ένα παράδειγμα. Το Nord Stream 2. Πέραν των προσπαθειών μας και μετά από τις συζητήσεις που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά από τις προσπάθειες που κάναμε για την εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου, το Nord Stream 2 είναι υποσυζήτηση, συνεχίζονται τεχνικές προετοιμασίες και υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες μπαίνουν στη σειρά για να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να παρουσιάσει το τελικό και πλήρες κείμενο της έκθεσής της για το Nord Stream 2 και για την εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου εξαιρέσει. Δεν πρέπει να συνεχιστεί το status quo σε ό,τι αφορά τις μεγάλες εταιρείε προσφοράς ενέργειας που είναι έτοιμες να διασπάσουν την ελληνική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από τα εμπορικά συμφέροντα, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες επιχειρήσεις, <clears throat> ακόμα και με την υποστήριξη των ε, κρατών μελών, προσπαθούν να διαλύσουν τη συνολική αντίληψη για μια ενεργειακή ένωση. Δεν πρέπει λοιπόν να υποβαθμίσουμε το επίπεδο της ρύθμισης και δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε και να υποτιμήσουμε τη σημασία της ασφάλειας προμήθειας με φυσικό αέριο. Ε, εκτιμώ λοιπόν ιδιαίτερα αυτή την έκθεση. Θα πρέπει να κάνουμε κάποτε μια συζήτηση, ίσως πιο τεχνικού χαρακτήρα, για να καταλάβουμε ποιο είναι ο αντίκτυπο αυτών των τεχνικών σημείων στα θέματα εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Α βρούμε την κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Η κυρία Θεοχάρου τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να εκφράσω κι εγώ την βαρέσκεια μου για την έκθεση. Νομίζω ότι καλύπτει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό αυτό που πρέπει να γίνει. Επισημένω δύο πολιτικές παραμέτρους οι οποίες δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη. Η μία είναι η αγωνιώδης προσπάθεια της Τουρκίας να μετατραπεί σε εναλλακτικό ενεργειακό ομφάλιο λόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό εμπεριέχει τους ίδιους κινδύνους που έχει και η παροχή μόνο από την Ρωσία, δηλαδή ε, η εκβιαστική διακοπή της ροής φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Τουρκία γνωρίζεται πάρα πολύ καλά πόσο εύκολο έχει το ζήτημα του εκβιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο ζητήματα ασφαλείας. Είναι μια χώρα εντελώς ανασφαλής με πάρα πολλές ε, πολεμικές ε, ε σειράξεις εν εξελίξει μέσα στην επικράτειά της υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι για την συνεχή επίθεση εναντίον των οποιονδήποτε αγωγών διέρχονται από την Τουρκία. Ε, ο δεύτερος παραγοντάς αφορά την παραγωγή φυσικού αερίου από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να επισυμβεί στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 30 χρόνια σε ποσοστό 30% και αν εμφανίζεται δύσκολη, που δεν είναι δύσκολη η μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγό από την Λεβαντίνη προς την Ρεβιθούσα κοντά στην Αθήνα, που είναι ο πρώτος σταθμός, μπορεί να γίνει η μεταφορά με, με ηλεκτρισμό, δεδομένου ότι είναι πολύ πρόσφατα που ψηφίσαμε το κονδύλιο των 2,5 δισεκατομμυρίων για την ενεργειακή ζεύξη Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και εφόσον η ροή μπορεί να γίνει από την Ευρώπη προς το Ισραήλ μπορεί να γίνει και ανάποδα. Η, το φυσικό αέριο του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Κύπρου μπορεί να καλύψει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Η Κύπρος δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι υφίσταται τη συνεχή πολεμική απειλή της Τουρκίας ότι εάν το επιχειρήσει θα ε, παρέμβει στρατιωτικά η Τουρκία. Λάβετε υπόψη και αυτούς τους παράγοντες και εμείς θα υποβάλουμε ε, τροπολογίες σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. σε ευχαριστούμε πολύ κυρία Θεοχάρους. Η κυρία Σουίτσα θέλει επίση το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρον το ότι συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα, τη στιγμή ακριβώ που ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος ε, Πούτιν συναντιόνται. Ενδιαφέρουσα αυτή η σύμπτωση. Υποστηρίζω πάντως την ε, γνωμοδότηση του συναδέλφου μας Σάριους Βόλσκι, αλλά έχω μία ερώτηση παρακαλώ, γιατί δεν ε, μου φαίνεται από τις τροπολογίες απάντηση. Για το 8 δισεκατομμύρια κυβικά που λέτε εσείς ότι πρέπει να αποτελεί το όριο. Πώς καταλήξατε σε αυτά τα 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Επίσης, είπατε ότι και τεχνικά πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία και η ρήτρα αλληλεγγύης. Γιατί αν μια χώρα εξαρτάται μόνο από έναν προμηθευτή, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και αλληλεγγύη. Εδώ έχουμε ένα πραγματικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Όσον αφορά τώρα τους κύριου παίκτε στην αγορά, δεν θα ήθελα να καταχραστούμε του ανταγωνισμού. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, για να επανέλθω το όριο των 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων που αναφέρεται στι τροπολογίες σας. Πάντως υποστηρίζω όλα όσα είπατε και έχετε γράψει και θεωρώ ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι αναγκαία, αλλιώς θα εξαρτώμεθα πάντα από την καλή θέληση των μεγάλων επιχειρήσεων φυσικού αερίου. Το ενεργειακό πρέπει να προχωρήσει και κατά τη γνώμη μου, όπως το είπατε κι εσείς, είναι αναγκαίο να επιδείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία. Η προσέγγιση μας πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη από ό,τι μέχρι τώρα. Στηρίζω λοιπόν την Επιτροπή και βασικά και τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σάριος Βόλσκι θα απαντήσει για το όριο αυτό των 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Παρακαλώ. μια μεγάλη σύμβαση την να πω, 55 BCM. Δισεκατομμύρια κυβικά. Τα δισεκατομμύρια δηλαδή κυβικά. Είναι κάτω από το 40% της γερμανικής ε, κατανάλωσης και δεν θα αναφέρεται. Κάθε μικρό συμβόλαιο όπως Λιθουανίας, Κροατίας, Λετωνίας, Εστονίας μικρές συμβάσεις δηλαδή, θα εκφράζονται σε ποσοστό. Οπότε, η μνήα στο μέγεθος της αγοράς θα είναι το κλειδί, ενώ θέλουμε να έχουμε μία αγορά φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, οι μικρές και μεσαίες θα αναφέρουν τις συμβάσεις τους και δεν θα αναφέρονται τα μεγάλα ε, συμβόλαια, τα οποία βέβαια σε σχέση με το μέγεθος ε, της αγοράς μιας χώρας μπορεί να θεωρούνται μικρά. Εγώ συμφωνώ και με την προσέγγιση του κύριου Ντέμεσμάκερ. Έχετε δίκιο ότι ο ανταγωνισμός είναι καλό σημείο αναφοράς. Οπότε θα συμφωνήσω με τις προτάσεις σας από αυτού. Αλλά υπάρχει και ένας παραλληλισμός εδώ. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, η DGCOM, ε, μπαίνει στο παιχνίδι κάθε φορά που γίνονται συγχωνεύσεις κλπ. πάνω από ε, κάποιο αριθμό δισεκατομμυρίων συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ε, την ίδια μεταχείριση. Αν πούμε λοιπόν 40% δεν θα αναφέρονται όλες οι συμβάσεις. Έχοντας μελετήσει διάφορες συμβάσεις πολλών χωρών συγκρίνοντας με Κατάρ, Νορβηγία, Ρωσία, Περού. Αυτό είναι το σωστό όριο. Μπορούμε να το συζητήσουμε. 5 ή 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αλλά το βασικό μου ερώτημα προς την Επιτροπή είναι ότι δεν πρέπει να τα μελετάτε όλα τα συμβόλαια αλλά είναι καλό να έχετε το δικαίωμα να μπορείτε να εξετάσετε όποια σύμβοση θέλετε, όποια στιγμή θέλετε. Γι' αυτό προτείνουμε το μέγεθος των συμβάσεων και όχι το ποσοστό, γιατί τότε μπαίνουν επίσης όρις όλες οι συμβάσεις. Η διαφάνεια των συμφωνιών μεταξύ κυβερνήσεων, που έχουν ήδη συμφωνηθεί δηλαδή από το Συμβούλιο, εντάξει. Αλλά των επιχειρήσεων είναι ακόμα πιο σημαντικές. Και όπως το είπατε και εσείς κυρία Σουίτς, υπάρχει όντως αυτή η σύμπτωση που συναντιούνται ο Γιούγκερ και ο Πούτιν σήμερα. Είναι αλήθεια ότι ο Γιούγκερ είναι αφοπλισμένος μπροστά στον Πούτιν. Ο Πούτιν τα ξέρει όλα. Είναι αυτός που λέει σε ποια τιμή και σε ποιον θα δώσει. Και ο Γιούγκερ δεν ξέρει τίποτα. Μόνο να μαντέψει μπορεί. Εμείς αυτήν την ασυμμετρία θέλουμε να την ξεπεράσουμε, γιατί είναι σε βάρος μας. Και θέλουμε επίσης να διορθώσουμε και αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή στην επιφάνεια υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις, αλλά στην πραγματικότητα όλα τα σημαντικά συμβόλαια είναι κρυμμένα. Ένα μέρος μόνο των συμβάσεων εμφανίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βάζει τις επιχειρήσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στη Δυτική Ευρώπη, σε άδικη θέση, σε μειονεκτική. Γιατί κάποιοι γνωρίζουν για τις συμβάσεις των ανταγωνιστών τους, ενώ άλλοι δεν γνωρίζουν. Οπότε πρόκειται για μια άδικη, ασύμετρη κατάσταση που δεν συνάδει με τον ακρογωνία ολίθο της οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι οι οικονομικοί φορείς όλοι μπαίνουν στο ίδιο επίπεδο, είναι ισότιμοι και τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε αυτό το 40% είναι πολύ πονηρό και δικαιολογείται μόνον εφόσον θέλουμε να δούμε κάποια μόνο συμβόλαια κάποιων ε, ενεργειακών εισίδων. Για μένα αυτή δεν είναι δικαιολογία. Και δεν πρέπει εδώ να αντιβαίνουμε στη φιλοσοφία την ενεργειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να ξεφεύγουν κάποιες συμφωνίες. Δεν μπορεί να κρύβεις κάποιες συμφωνίες και να εμφανίζεις κάποιες άλλες. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση αυτή. Θυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ποια είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες αύριο το μεσημέρι. Περνάμε στο σημείο 10. Θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά διακυβερνητικέ συμφωνίε και μη δεσμευτικά μέτρα μεταξύ 100 μελών και τρίτων χωρών στον τομέα τη ενέργεια και κατάργηση της απόφασης 994 2012 ΕΕ. Η μας εδώ είναι ο Έδουαρτ Κούκαν και η αρμόδια επιτροπή είναι η ΙΤΡΕ. Έχουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότησης και είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Κούκαν για να παρουσιάσει το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Αντρέ. Η γνωμοδότηση αυτή ακολουθεί την πρόταση της Κομισιόν για μια απόφαση η οποία επικαιροποιεί το μηχανισμό λήψης απόφαση ορισμένε διακυβερνητικές αποφάσεις στο, συμφωνία στον τομέα της ενέργειας. Είναι ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Η γνωμοδότησή μου λέει ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι λογική και αυτή γραμμίζεται με τη θέση του Κοινοβουλίου που ενεκρίθη πέρσι το Δεκέμβριο για τη στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης. Στην έκθεση αυτή ζητήσαμε μια πιο στεναρή στάση της Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις για τις διακυβερνητικές συμφωνίες και που να συμπεριλαμβάνει μια εκ των προτέρων αξιολόγηση της ε, συμφωνίας προτού υπογραφεί η συμφωνία με την τωρινή νομοθεσία. Όταν η Κομισιόν κάνει εκ των υστέρων εξ αναλύσεις των διακυβερνητικών συμφωνιών είδαμε ότι η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να φέρει όλες αυτές τις προβληματικές συμφωνίες να τις ευθυγραμμίσει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί για να μπορούμε να έχουμε μια λειτουργική ενεργειακή ένωση. Για τις λεπτομέρειες τώρα της πρότασης Κομισιόν. Η εμβέλεια της τωρινής πρότασης καλύπτει όχι μόνο διακυβερνητικές συμφωνίες, αλλά και μη δεσμευτικές νομικές συμφωνίες. Μπορεί να υπάρχουν μνημόνια ε, κατανόησης, συναντήληψης ή πολιτικές δηλώσεις. Δεν καλύπτει βέβαια τι εμπορικέ συμφωνίε μεταξύ επιχείρησεων που είναι σε, άλλη, σε άλλο πλαίσιο. Συμφωνώ με τα κύρια σημεία λοιπόν τη πρόταση Κομισιόν ότι παραδείγματος τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρούν ενήμερη την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την έναρξη διακυβερνητικών συζητήσεων και σε ό,τι αφορά την, πρόταση, την πρόοδό του. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Κομισιόν για αξιολόγηση κατά πόσο συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο πρώτου υπογραφούν. Τα κάτι μελη θα πρέπει να πληροφώνουν την Κομισιόν για μη δεσμευτικού χαρακτήρα ενεργειακέ συμφωνίε με τρίτες χώρε. Και η δική μου πρόταση είναι καταρχήν να υπογραμμίσω δύο θέματα. Θέλω να υπογραμμίσω θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μένα για να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για τις συμφωνίες αυτές, να φέρουμε περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και περισσότερη διαφάνεια στον τομέα των συμφωνιών σε ενεργειακά θέματα και παράλληλα η Κομισιόν πρέπει να εξασφαλίσει την διαφύλαξη του απορρίπτου σε αυτές τις συμφωνίες. Επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να δει κατά πόσο συμμορφώνονται αυτές οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, λαμβάνοντας όμως και υπόψη την στρατηγική ασφάλειας στα ενεργειακά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω λοιπόν τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας για την γνωμοδότηση αυτή. Οι τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν μέχρι αύριο το μεσημέρι. Έχετε 25,5 λοιπόν ώρες για να καταθέσετε Σε Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Έντβαρτ, λέει ο Πρόεδρος. Α, παντού. Παντού βλέπω τον κύριο Πιτζουλα, γιατί παντού είναι σκιώδης εισηγητής. Βγαίνω, βγαίνω από τις σκιές ως σκιώδης και έρχομαι στο προσκήνιο, στο φως. Συνεχίζω στα κροατικά, πρόεδρε. Έχω να επισημάνω τρία βασικά προβλήματα. δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος των προτέρων, η δυνατότητα συμμετοχής διπλωματεύσης και επίσης δεν έχουμε κάποιον ε, ε, μηχανισμό ακύρωσης αυτών των συμφωνιών. Οπότε δεν υπάρχει διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Η απόφαση αυτή δεν ε, μας δίνει περιθώριο εναρμόνισης των όσων αφορούν σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης το να έχουμε αυτού του είδους της συμμόρφωσης εκ των υστέρων σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση των συμβάσεων. Άρα θα πρέπει να τροποποιηθεί αυτή η απόφαση. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει συνένεση. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια επαρκή ανταλλαγή πληροφοριών και υπάρχουν εγγυήσει για ασφαλεία δικαίου, αν επομένως υπάρχουν κάποιες διατάξεις συμβάσεων που αντιβαίνουν στο κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει ε, να εκδώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης θα πρέπει να επαρρυπνεί ούτω ώστε να υπάρχουν και να τηρούνται οι προθεσμίες των διαπραγματεύσεων και έτσι να εξασφαλιστεί η ενεργειακή μας ασφάλεια. Άρα χρειάζεται περισσότερη ε, διαφάνεια όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών ε, εφοδιασμού και ανεφοδιασμού Χρειάζεται επομένω να πετύχουμε τον στόχο μας, να θέλουμε, να συνάδει η εμπορική πολιτική με την εξωτερική μας πολιτική και να αναγνωρίσουμε ότι λόγω των εισαγωγών ενεργείας θα πρέπει έτσι να δούμε τη συμβάση με τα ε, τρίτα μέρη, με τους τρίτες χώρες. Άρα θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικότητα στην ε, ε, ενέργεια και να αποκτήσουμε κάποια αυτονομία. Σας ευχαριστούμε. Λέω πρώτος, θέλει κάποιο το λόγο. Επ' αυτού δεν βλέπω να ενδιαφέρει να λάβει το λόγο για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, Έντουερτ. Α, Σάριος Βόλσκης το λόγο. Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρθηκαν και παρατηρώ το εξής οι διακυβερνητικές συμφωνίες είναι εκείνες που προηγούνται των συμβάσεων των εταιριών. Επομένως, πάμε σε αυτά που σας παρουσίασα εγώ προηγουμένως. Δηλαδή, αυτά που σας είπα εγώ συμπληρώνω αυτά που είπε ο Έντουαρτ Κούκαν. Όσο πιο ξεκάθαρε είναι οι συμφωνίες οι τόσο λιγότερα προβλήματα γεννώνται αργότερα όσον αφορά τα μυστικά deal των εταιριών. Δεν υπάρχουν ε, συμβόλαια που δεν επηρεάζονται από την πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Ίσως μια μέρα να γίνει αυτό. Αλλά προς το παρόν όλα είναι χρωματισμένα πολιτικά. Και υπάρχει και ε, πάντοτε μια μεταβλητή γεωπολιτική. Έφυγε ο Πέτρας. Δεν πρόκειται όμω για καθαρά εμπορικό χαρακτήρα σύμβασης. Όσο πιο σαφή είναι τη διακυβερνητικά σύμφωνα τόσο καλύτερα. Και επομένω θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε τις αρνητικές συνέπειες. Όπως ε, την αμφισβήτηση ε, της σύμβασης της Βουλγαρίας ε, με την Gazprom για το South Stream. Και ίσως θα πρέπει επομένως να έχουμε πρόληψη των καταστάσεων αυτών με τέτοιο έλεγχο επί των ε, συμφωνιών και να αποφύγουμε επομένω καταστάσεις τέτοιες και για κάποιες ε, συμφωνίες που δεν είναι ε, ονομαστικά, δεν είναι θεωρητικά διακυβερνητικές. Αυτά τα μνημόνια, τα οποία ουσιαστικά έχουν διακυβερνητικό χαρακτήρα και είναι ε, ακόμα πιο σημαντικά τα μνημόνια από τις ε, επίσημα διακυβερνητικές διακρατικές συμφωνίες. Γι' αυτό σας λέω, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει όπως και να χαρακτηρίζονται νομικά οι συμφωνίες ε, των κυβερνήσεων θα πρέπει να διέπονται από σαφήνεια και διαφάνεια. Θέλετε να ε, συνοψίσετε συγκεκριτά ο κύριος Κούκαν. Μόνο μια φράση ευχαριστώ τον ε, Σάριους Βόλσκε και είναι ε, σαφές το ότι όταν έχουμε ε, ξεκάθαρες διακυβερνητικέ συμφωνίες τόσο καλύτερες είναι οι εξελίξεις για τις συμφωνίες που ακολουθούν και επίσης αυτές οι διακυβερνητικέ συμφωνίες όπως και τα διάφορα μνημόνια και δηλώσεις επίσημες καλύπτονται από αυτό το οποίο προτείνω ως μηχανισμό που θα επιβάλλει τη διαφάνεια και τη σαφήνεια. Ευχαριστώ, Έντουαρτ, λέει ο κύριος Πλέγκοβιτς. Εδώ λιγώνεται η συζήτηση για το 10. Αύριο θα ψηφίσουμε, και, μάλλον αύριο, λίγη προθεσμία κατάσταση των τροπολογιών 15 Ιουνίου το μεσημέρι. Η συνέχεια της συνεδρίας θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, επομένως επιβάλλεται μια διακοπή δεκάλεπτη. Θα έρθει η κυρία Νατάλια Αποστόλοβα, νεοδιοριστής επικεφαλής της αντιπροσωπείας στο Κωσυφοπέδιο θα έρθει για συζήτηση. Οπότε, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν επιτρέπεται να παρίστανται σε συνδυάσει και κλεισμένων, παρακαλώ κατά τη διάρκεια της δεκάλεπτης διακοπής, να εγκαταλείψουν την αίθουσα και να έρθουν στις 11.30 ε, περίπου τότε που θα έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον Σαραχαδίν Ντεμίρτα, τον συμπρόεδρο του Δημοκρατικού Λαϊκού κόμματο της ε, Τουρκίας, που με εκείνο το θέμα θα ολοκληρώσουμε τα πρωινά μα σημερινά θέματα. Αλλά 10.45 θα έχουμε την ε, ε, επικεφαλής αντιπροσωπεία για το Κόσοβο. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε την ε, ημερησία διαταξή μας. Έχουμε την ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, συμπρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, ΧΑΝΤΕΠΕ. Θέλω καταρχήν να καλωσορίσω τον κύριο Ντεμιρτάς εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, μαζί με τους συνεργάτες του. Ο κύριος Ντεμιρτάς Γνωρίζετε, κύριε Δημητά, ξέρετε ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βρέθηκε και στη μέση διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακολουθούμε όλοι από πολύ κοντά την κατάσταση στην Τουρκία, τόσο σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας, τα θέματα πολιτικής εξέλιξης, την κρίση μετανάστευσης και προσφύγων τα εξωτερικά λοιπόν αυτά θέματα, αλλά και τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα ακούσουμε σήμερα τη δική σας ανάλυση της κατάστασης στην Τουρκία σήμερα. Η μεγάλη τουρκική εθνοσύνελευση έχει ψηφίσει μια τροπολογία στο τουρκικό σύνταγμα που επιτρέπει την ε, άρση της ασυλίας βουλευτών της ε, συνέλευσης και την προηγούμενη εβδομάδα οι ευρωβουλευτές έγιναν το ανάστημά του για να καταδικάσουν αυτή την πράξη πολιτικής πίεσης και ο Επίτροπος Χάν εξέφρασε την ανησυχία του για τις ανησυχητικές αυτές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τη δική σας ανάλυση, τις δικές σας απόψεις, ώστε να εμπλουτίσουμε τις πηγές πληροφόρησης και ανάλυσης για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση της Τουρκίας και το γενικό πλαίσιο του διαλόγου Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο των αποφάσεων σε σχέση με την <clears throat> φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων και τη συνέχιση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας και το συνολικό φυσικά πλαίσιο της επίτευξης μιας λύσης για, ε, για τον έλεγχο των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά και την κατάσταση των Κούρδων στην Τουρκία Έχετε περίπου 10-12 λεπτά για τις αρχικές σας παρατηρήσεις, κύριε Ντεμετάς, και μετά θα ακολουθήσουν τα σχόλια των βουλευτών και θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε πάλι στο τέλος για 10 λεπτά περίπου. 25 είναι το κανάλι της τουρκικής γλώσσας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να εκφραστώ ενώπιόν σας. Ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προφανώς παρακολουθείτε από πολύ κοντά τις εξελίξεις στην Τουρκία και είμαι σίγουρος ότι έχετε λεπτομερείς πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να μοιραστώ τις απόψεις μου μαζί σας σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία και άλλες εξελίξεις και γεγονότα που μπορεί να επισυμβούν στο μέλλον. Η Τουρκία περνάει αυτή τη στιγμή μια εξαιρετικού χαρακτήρα πολιτική κατάσταση. Αυτό δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση γιατί το Σύνταγμα είναι σε αναστολή. Εμποδίζονται οι εκφράσεις κάθε ελευθερίας. Τα δικαιώματα των πολιτών, τα συνταγματικά δικαιώματα παραβιάζονται κάθε μέρα όλο και περισσότερο οικοδομείται ένα μονοκομματικό κράτος υπό την ηγεσία του Ταγί Περτογάν. Φυσικά υπάρχουν ιστορικοί λόγοι για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Τα προβλήματα αυτά δεν δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός. Έχουμε σοβαρά προβλήματα δημοκρατίας από την αρχή της τουρκικής δημοκρατίας. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να αποδοθούν σε σφάλματα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν όμως και η κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ δεν έχουν κάνει τίποτα για να εισαγάγουν μεταρρυθμίσεις και να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, έχουν δημιουργήσει περισσότερα και πιο πολύπλοκα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την διαδικασία ειρήνευση, η οποία κράτησε για ε, περισσότερο από δύο χρόνια και ανεστάλλει σταμάτησε η κατάπαυση του πυρός διότι ο κύριος Ερδογάν θεώρησαν ότι, θεώρησαν ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγούσε σε απώλεια ψήφων στις εκλογές πέρσι της 7η Ιουνίου. Επομένως σταμάτησε την όλη διαδικασία ειρήνευσης στην νοτιοανατολική Τουρκία και ακολούθησαν αναζωπηρώσεις των ε, αντιπαραθέσεων. Υπήρξε μια κατάσταση ε, ολέθρου σε πολλές περιοχές της ε, νοτιοανατολικής Τουρκίας. Υπάρχουν περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας εδώ και έξι μήνες, όπου γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις με άρματα μάχης. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ισοπεδωθεί. Περίπου 500.000 άτομα έχουν ε, αναγκαστεί να φύγουν από τις αιστείες τους. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν φωνευτεί σε αυτές τις εχθροπραξίες και μαχητές του ΠΚΚ και δυνάμεις ασφαλείας αλλά και πάρα πολλοί άμαχοι ο Ερντογάν αρνείται να κάτσει σε τράπεζα διαπραγματεύσεων για να υπάρξει λύση όμως στο πρόβλημα αυτό. Η αντιπαράθεση αυτή τον ευνοεί, ευνοεί τους πολιτικούς στόχους τους. Ο πόλεμος ο οποίος γίνεται στην Ανατολική Τουρκία ουσιαστικά τροφοδοτεί εθνικιστικά συναισθήματα και επομένως ο Ερδογάν ευνοείται από τα εθνικιστικά και πατριωτικά αυτά συναισθήματα και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει να προχωρήσει σε επανέναρξη της ε, διαδικασίας ειρήνευσης. Η άρση της ασυλίας των βουλευτών επίσης είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα χωριστά. Είναι τμήμα της στρατηγικής του Ερδογάν. Ήρθαν οι ασυλίες πολλών από τους βουλευτές μας σε παραβίαση του, συντάγματο. του συντάγματος. Υπάρχει ένα πρόσθετο άρθρο σε αυτή την τροπολογία το οποίο περιορίζει το δικαίωμά μας να έχουμε προσωπική προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο. Επομένως, μια αντισυνταγματική τροπολογία έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μας και το τελευταίο άρθρο αυτής της τροπολογίας μας εμποδίζει να κάνουμε ως άτομα <clears throat> προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας. Οι φάκελοι των ερευνών για τους βουλευτές του ΧΑΝΤΕΠΕ είναι περίπου 600 τέτοιοι φάκελοι. Εγώ έχω 93 έρευνες εναντίον μου με τις οποίες εγώ μπορώ να διωχθώ και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει ήδη την επόμενη εβδομάδα η δίωξη εναντίον μου. Το Υπουργείο με Δικαιοσύνη έχει δώσει στους αρμόδιους εισαγγελεί του φακέλου αυτού και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίωξη την επόμενη εβδομάδα. Η ομάδα μα, το κόμμα μα, αποφάσισε να μην ανταποκριθεί στις προσκλήσεις των εισαγγελέων. Δεν θα δεχτούμε να καταθέσουμε δεν θα δεχτούμε να κάνουμε δηλώσεις γιατί θεωρούμε ότι η άση της ασυλίας μας αποτελεί μια παραβίαση του τουρκικού <clears throat> συντάγματος. Και όλοι οι εισαγγελείς εργάζονται με, εκτελώντας εντολές του Ερντογάν. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν οι εισαγγελείς να μας σύρουν ενώπιον του δικαστηρίου δια της βίας. Όταν γίνει κάτι τέτοιο όμως με χρήση βίας εμείς δεν θα ανταποκριθούμε στα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν από το δικαστήριο και έχουμε ένα κείμενο, ένα κοινό κείμενο υπεράσπισης. Όλοι οι βουλευτές δεν θα κάνουμε νομική υπεράσπιση, θα τονίσουμε απλώς ότι πρόκειται για μια πολιτική δίωξη η οποία στοχεύει στο να οικοδομήσει το μονοκομματικό κράτος στην Τουρκία. Δεν θα απαντήσουμε σε κανένα από τα ερωτήματα που θα τεθούν από εμά σε εμά από τους εισαγγελείς. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν θα βρεθούμε στη συνέχεια στη φυλακή. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι φάκελοι έρευνα εναντίον μας, οι οποίοι είναι κομικοτραγικοί. Οι περισσότερες έρευνες που αφορούν τους βουλευτές του ΧΑΝΤΕΠΕ έχουν να κάνουν με ελευθερία έκφρασης. Εγώ έχω τρει τέτοιες περιπτώσεις φακέλους ανακριτικούς εναντίον μου που έχουν να κάνουν με ομιλίες και δηλώσεις που έχω κάνει μέχρι σήμερα Έχω κοιτάξει τους φακέλους αυτούς, έχω δει τις ε, κατηγορίες εναντίον του εαυτού μου και από νομική άποψη είναι πραγματικά ικτρές. Το 2008, παραδείγματος χάρη, στις, ε, στην ε, εορτασμό του Ναυρούς της κουρδικής πρωτο, πρωτοχρονιάς, είπα το εξή. και κατηγορούμε ως ότι έκανα προπαγάνδα υπέρ ενός τρομοκρατικού, τρομοκρατικής οργάνωσης. Είπα το εξή ότι ο πιο σύντομος δρόμος για την ειρήνη περνάει από τον κύριο Ελτζαλάν. Είναι ο συντομότερος και ο λιγότερο αιματηρός ε, δρόμος ειρήνης. Εμείς αγωνιζόμαστε για την αδελφότητα και την ειρήνη για πολλά χρόνια. Δεν θέλουμε περαιτέρω αιματοχυσία, θέλουμε διάλογο οι Κούρδοι. Και οι Τούρκοι δεν αξίζει να νιώθουν το σημερινό πόνο που νιώθουν. Αυτό θεωρείται ότι είναι προπαγάνδα υπέρ μια τρομοκρατική οργάνωση και με κατηγορούν. Αυτή είναι μία από τι κατηγορίε που εκκρεμούν εναντίον μου. Μια, άλλο παράδειγμα. Σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, στην Κεσάρια, το κτίριο του ΧΑΝΤΕΠΕ έτυχε επιθέσεων από ρατσιστικές δυνάμεις. Κάηκε, καταστράφηκε και εμείς καταθέσαμε μία ε, αγωγή εναντίον της αστυνομίας στην πόλη της Κεσάριας, λέγοντας ότι έδειξε αμέλεια ότι δεν προστάτευσε το κτίριό μας μετά από την προσφυγή αυτή, ο εισαγγελέα άρχισε μία δίωξη εναντίον μας για προσβολή και συκοφαντία του, της αστυνομικής αρχής. Αντί λοιπόν να ερευνήσει την αδράνεια της αστυνομίας, εμείς θα κατηγορηθούμε για ε, δυσφήμιση των αστυνομικών δυνάμεων στην Κεσάρια. Μία άλλη κατηγορία εναντίον μας σε μια προεκλογική συγκέντρωση έκανα μια ομιλία στα κουρδικά που είναι η δική μου γλώσσα. Ο εισαγγελέα δεν έχει κανένα πρόβλημα με το περιεχόμενο της ομιλίας, θεωρεί όμως ότι είναι αδίκημα το ότι χρησιμοποίησα την κουρδική γλώσσα. Και υπάρχει έρευνα που εκκρεμεί εναντίον μου. Τέσσερις, τέτοιες, τέσσερις τέτοιοι φάκελοι υπάρχουν εναντίον μου για το γεγονός ότι έχω χρησιμοποιήσει την κουρδική γλώσσα. Εγώ είπα ότι ο, λαός του, ο κουρδικός λαός έχει το δικαίωμα να έχουν σχολική παιδεία στα κουρδικά. Και αυτό τώρα είναι αντικείμενο ε, κατηγορίας εναντίον μου. Όλοι λοιπόν αυτοί οι φάκελοι έχουν να κάνουν με θέματα ελευθερίας έκφρασης. Όλοι οι βουλευτές μας κατηγορούνται γιατί έχουν μιλήσει ελεύθερα και έχουν εκφράσει τις απόψεις τους. Είναι πραγματικά ντροπή ότι γίνεται αυτή η δίωξη εναντίον μας και κινδυνεύουμε να βρεθούμε στη φυλακή. Και εγώ αυτή τη στιγμή έχω να επικρέμονται πάνω μου 465 χρόνια φυλάξης αν εγκριθούν όλες αυτές οι διώξεις και καταδικαστώ. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν ο Ερντογάν να περάσει κάτι τέτοιο. Ήταν εύκολο να το περάσει αυτό από το Κοινοβούλιο και μετά από αυτό θα έχει πια μια μόνο προσωπική εξουσία. Το να υπάρχουν Κούρδοι βουλευτές στην μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση είναι κρίσιμο χαρακτήρα. Γιατί εμείς είμαστε η μόνη ανασχετική δύναμη η οποία μπορεί να σταματήσει τον κύριο Ερντογάν. Πετάμε λοιπόν μια ιστορική στιγμή για το μέλλον της Τουρκίας. Μέσα σε αυτή την χρονική στιγμή πιστεύουμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιτύχουν την ειρήνη στην Τουρκία πρέπει να ενισχυθούν για να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα μας. Και αυτό είναι απαραίτητο για την ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα μας για να επιτευχθεί και η ειρήνη και η σταθερότητα στη Συρία. Γιατί είναι προϋπόθεση η ειρήνη και η σταθερότητα στην Τουρκία. Να υπάρξει μια συμφιλίωση Τούρκων και Κούρδων αυτό θα μπορέσει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στη Συρία. Έχουμε όλοι μας την πρόκληση της κρίσης της προσφυγική. Η ειρήνη μεταξύ Κούρδων και Τούρκων θα έχει μεγάλη επιρροή στην επίλυση του προσφυγικού προβλήματος. Θα υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον στην ε, ε, νοτιοανατολική Τουρκία και την Ρόζαβα, το, την περιοχή της Συρίας που ελέγχεται από τους Κούρδους, αλλά ο Ερντογάν δεν θέλει να συμφιλειωθεί με τους Κούρδους της Συρία και γι' αυτό συνεχίζεται η αστάθεια. Στο βόρειο τμήμα όμως της Συρίας υπάρχει σταθερότητα που μπορεί να επιτευχθεί πολύ γρήγορα και αν γίνει κάτι τέτοιο θα μπορέσουν οι περισσότεροι από τους Σύριους πρόσφυγες να επανέλθουν στις αιστείες τους γιατί θα υπάρχει μια ασφαλής περιοχή για αυτούς τους ανθρώπου στη Συρία. Θα είναι σε θέση να επανέλθουν στις αιστείες τους. Οι κουρδικές αρχές στη Ροζάβα συνεργάζονται και έχουν δείξει τη θέληση να ε, υποδεχτούν όλους τους ε, πρόσφυγες από την περιοχή αυτή, είτε είναι Κούρδοι είτε έρχονται από άλλη εθνοτική ομάδα. Επί τη βάση λοιπόν του προβλήματος αυτού του προσφυγικού θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτό είναι αλληλένδετο με την διαδικασία ειρήνευσης στην Τουρκία. Αν δεν γίνει τίποτα σε σχέση με την ε, αντιπαράθεση που σοβεί ακόμα στην Τουρκία, οποιαδήποτε λύση στη Συρία θα είναι μονάχα προσωρινή. Ο Ερδογάν αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί την κρίση των προσφύγων ως ε, μέσο εκδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικές πολιτικές για να εμποδίσουμε αυτή τη ε, διαδικασία. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξετε τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Τουρκία και η εσωτερική διαδικασία ειρήνευση στην Τουρκία θα πρέπει να επανεκκίνησει και να υπάρξει υποστήριξη προς την διαδικασία αυτή και επίσης οι περιοχές που βρίσκονται στην Βόρεια Συρία και έχουν κουρδική ηγεσία, θα πρέπει να ενισχυθούν. Αν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, κάποια από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να επιληθούν. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει με πιο αποφασιστικό τρόπο και να παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, παραγωγικά να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή για την επίλυση του, του κουρδικού προβλήματος στην Τουρκία, αν μπορέσει να πάει μια αντιπροσωπεία διαμεσολάβησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν μπορείτε να πάρετε λοιπόν πιο έντονα και πιο συγκεκριμένα βήματα για τα θέματα αυτά, θα μας διευκολύνεται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να αναζωογονηθεί η διαδικασία ειρήνευσης. Μπορεί την άλλη εβδομάδα και εγώ και οι συνάδελφοί μου να βρισκόμαστε στη φυλακή. Θα χρειαστούμε λοιπόν την υποστήριξή σας, την αλληλεγγύη μας, την αλληλεγγύη σας. Εμείς δεν θα φύγουμε από τη χώρα μας. Θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο να μας φυλακίσουν να μας φυλακίσουν ακόμα και για χρόνια, αλλά δεν θα φύγουμε από τη χώρα μας, γιατί ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την ειρήνη στη χώρα μας. Αν υπάρξει διεθνής υποστήριξη, αν υπάρξει διεθνής αλληλεγγύη, θα υπάρξει και μια εύθερη ευκαιρία για μας να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στην Τουρκία. Και αυτό θα είναι και ένας τρόπος να προωθήσουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία. Θα υπάρξουν προβλήματα μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ερντογάν έκανε χθε μια ομιλία όπου είπε ότι θα επανεξετάσει το θέμα της συμφωνίας με την Ευρώπη και στο φως των επικρίσεων που διατυπώθηκαν από την Ευρώπη μπορεί να, ανα, να αναστείλει όλα αυτά τα θέματα. Μα αυτό δεν είναι ένα πολιτικό θέμα. Αυτό είναι μια διακυβερνητική υπόθεση. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ο Ερντογάν ο οποίο αποφασίζει μονομερό να σταματήσει τι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα διαπραγματεύσεων η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά. Χάρη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις εσείς έχετε κάποιο μοχλό πίεσης στην Τουρκία. Μπορείτε να μας βοηθήσετε αν κλείσουν τελείως όμως οι πόρτες και δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι και σε βάρος της δημοκρατίας. Πρέπει όμως να διατηρηθεί η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα ζητώντας το σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεχάγης και των ευρωπαϊκών αξιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ και τώρα μπορώ να ακούσω τα σχόλια και τις ερωτήσεις σα. Thank you ευχαριστούμε κύριε Ντιμετάς, λέει ο Πρόεδρος. Ε, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζει ο κύριος Πλέγκοβιτς, πριν αρχίσουμε την συζήτηση, παρακαλώ για την κατανόηση και συνεργασία σας. Σχεδόν 15 συναδελφοί μου ζητήσει τον λόγο. Άρα ο καθένα πρέπει να μιλήσει ένα λεπτό. Παρακαλώ τηρήστε αυτό το όριο, ούτω ώστε να επιτραπεί σε όλους τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο και να απευθυνθούν στον κύριο Ντεμιρτά. Κύριε Πύρη που είναι η συγκεκριά μας, κατόπιν τον κύριο Κεφαλογιάννη, επικεφαλή αντιπροσωπεία και εσεί αν θέλετε λάβετε το λόγο. Δεν θέλετε. Όχι, όχι, όχι τώρα κύριε Κεφαλογέννη. Πετε μου αν θέλετε να, να λάβετε το λόγο. Ναι, λέει ο κύριο Κεφαλογέννη μετά. Κυρία Πύρη, λοιπόν, που είναι η συγκέντρια, κατόπιν επικεφαλή τη αντιπροσωπεία, ο κύριο Κεφαλογέννη. Ε, ας προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το όριο. Ευχαριστούμε και την Τέμερτα που ήρθατε και μα δώσετε την ευκαιρία να σα ακούσουμε, ζητήσατε αλληλεγγύη. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο επέκρινε πάρα πολύ αυστηρά αυτά τα οποία γίνανε στην Τουρκία, δηλαδή για την άρση τη ασυλία τόσων βουλευτών, αλλά γνωρίζουμε ότι το ΧΑΝΤΕΠΕ είναι ο στόχος και αν ε, εξαφανιστείτε από το Κοινοβούλιο και βρίσκεστε πίσω από τα κάγκελα, εμείς ουδέποτε θα δώσουμε το πράσινο φως στην κατάργηση της θεώρησης διαβατηρίου. Ε, επομένως, ε, υπάρχει αλληλεγγύη, θα συνεχίσει να ισχύσει η αλληλεγγύη και θα είμαστε υπέρ ε, των βουλευτών που έχουν το δικαίωμα του λόγου. Ακόμα και εάν δεν συμφωνούμε με όσα έχετε να πείτε, ιδίω για ένα κοινοβούλιο ισχύει αυτό. Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά ε, το ανατολικό τμήμα της χώρας. Πέστε μας δύο λόγια για το τι γίνεται σε αυτές τις ε, πόλεις που υπάρχει απογόρευση κυκλοφορίας, τι γίνεται με του εκτοπισμένους και επίσης κάτι άλλο. Υπάρχει εδώ ευρεία πλειοψηφία που θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται με τίποτε η βία, δεν δικαιολογούνται με τίποτε οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Ξέρω ότι συμφωνείτε με αυτό το επιχείρημα, αλλά για πέστε μας, ε, εσείς τι κάνετε για να πείσετε το ΠΚΚ να καταθέσει τα όπλα. Ένα λεπτό κύριο Κεφαλογέννης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να καλωσορίσω και τον κύριο Δημητρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά να ρωτήσω πώ θα κατάφερε και ήρθε εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι ε, υποδιωγμού και ο ίδιο. Και θα ήθελα να ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοί του από το κόμμα του μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μα πληροφορήσουν για τα θέματα αυτά. Θέλω επίση να σημειώσω το μετριοπαθή λόγο του, νομίζω ότι βοηθάει προ την κατεύθυνση να έχουμε μια σταθερή Τουρκία, Τουρκία τη θέλουμε να παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή και αυτό βγαίνει και από το δικό του λόγο. Συνεργασία και συζήτηση και διάλογος πρέπει να υπάρξει από τη μεριά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την έκθεση την οποία ψηφίσαμε και στην τελευταία Ολομέλεια ε, για, τις, για, τους, για, τη, για τους διωγμούς των 153 βουλευτών ε, όλα τα, όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν σαφή και συγκεκριμένη θέση. Θέλω να ενημερώσω επίση, κύριε Πρόεδρε, <clears throat> την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι βρίσκουμε τεράστιε δυσκολίε για συνεργασία για την ε, μειχτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία με του συναδέλφου μα από, το, από το Τουρκικό Κοινοβούλιο. Ήδη έχει αναλάβει πρωτοβουλίε ε, και ο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν δύο αποστολέ, οι οποίε οργανώνουμε για το επόμενο διάστημα για τον Ιούλιο. Εμεί θα κάνουμε από τη μεριά του Κοινοβουλίου ότι μπορούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση δηλαδή η Τουρκία να μείνει σταθερή και να υπηρετήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και του δημοκρατικού θεσμού σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Thank Εμεί ευχαριστούμε, κύριε Κεφαλογιάννη, λέει ο Πρόεδρο. Εντάξει με την μετάφραση. Ναι, ακούτε τη μετάφραση. Όχι, όχι, δεν ακούσαμε. Μπορείτε να ελέγξετε με τον τεχνικό. Όχι, όχι, ο κ. Δημιρτάς. Δεν μπόρεσα να ακούσω τη μετάφραση από τον προηγούμενο μιλητή. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί δεν μπόρεσα να ακούσω τη μετάφραση. Εννοείται τον κύριο Κεφαλογιάννη, δεν ακούσατε από μετάφραση. Ναι, ναι. Παρακαλώ παραλάβετε αλλά συνοπτικά. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Δημητρά. Ε, το ερώτημά μου ήταν ε, πώ κατάφερε και ήρθε εδώ, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι υποδιώμο, γιατί θέλουμε και άλλα στελέχη και από το κόμμα του και από αυτού οι οποίοι διώκονται να, να έρχονται στο κοινοβούλιο και να μα ενημερώνουν. Θέλουμε μια Τουρκία σταθερή. Ε, χαίρομαι γιατί ο λόγο του είναι μετριοπαθή και αυτό βοηθάει τον διάλογο και τη συνεργασία που χρειάζεται να υπάρχει στην Τουρκία ώστε ένα παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτή την Ολομέλεια αλλά και στην έκθεση την οποία ψηφίσαμε έχει δείξει ότι ε, αγωνίζεται προς την κατεύθυνση των δημοκρατικών θεσμών και την προστασία των, των μειονοτήτων. Επίσης ε, ενημέρωσα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ότι βρίσκομαι τεράστιες δυσκολίες για να προχωρήσω με τη συνεργασία στην Μιχτή Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, διότι βρίσκομαι ε, μια δυσκολία συνεργασίας με τους συναδέλφους μας από το Τουρκικό Κοινοβούλιο οι οποίοι φαίνεται ότι σε αυτή, το, σε αυτή την περίοδο που γίνονται μεγάλες αλλαγές όχι προς δημοκρατική κατεύθυνση με την αλλαγή του συντάγματος δεν συνεργάζονται όπως εμείς θα θέλαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, κύριε Γκόπες. Όχι. Η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ δύσκολο για μας. Έχουμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία από τη μια, που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε πιεστεί πολύ με το μεταναστευτικό. Από την άλλη μεριά Θέλουμε να βοηθήσουμε την αντιπολίτευση στην Τουρκία γιατί η κατάσταση είναι αφόρητη. Και με όλα αυτά που έχει κάνει ο κύριος Ντοργάνο, οπότε τι μας προτείνεται να κάνουμε. Πρέπει να σταματήσουμε τις διαπραγματεύσει για προσχώρηση της Τουρκίας, να σταματήσουμε να μιλάμε, να σταματήσουν όλα. Ο πρόεδρος κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι η Τουρκία κάνει βήματα πίσω αντί για μπροστά. Και επομένως πάρα πολλοί από τους συναδέλφους μας βρίσκονται σε κατάσταση ακατανοησίας. Εμείς δεν μπορούμε ως Κοινοβούλιο να είμαστε διπλωματικοί σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να πούμε σαφώς την άποψή μας. Δεν είμαστε διπλωμάτες, δεν είμαστε εκπρόσωποι χωρών. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την τήρηση των κριτηρίων Όπω είπε η Κατυπήρη, δεν μπορούμε εμεί να συμφωνήσουμε για τη φιλελευθερωποίηση των προξενικών θεωρήσεων κατά τέτοιε Ο κύριο Λόπε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι η επίσκεψη αυτή θα βοηθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση της προσωπικότητάς σας και του κόμματός σας και του ρόλου που παίξατε στη διαδικασία ειρήνευσης ε, στην Τουρκία και φυσικά υπάρχει απόλυτη αλληλεγγύη από τη δική μας πλευρά για τους βουλευτές της, ε, του κόμματός σας και αυτό το οποίο περνάνε τώρα. Μιλήσατε για την κατάσταση που περνάει ο κουρδικό λάο και τον πόλεμο που έλαβε χώρα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Θα ήθελα όμω μερικά πιο συγκεκριμένα στοιχεία, όπω η, η κρίση σα για την Συμφωνία ευρωπαικη Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία που συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο μα τι τελευταίε ε, εβδομάδε. Εμεί έχουμε επικρίνει πάρα πολύ τι αυταρχικέ τάσει του Ερδογάν, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε ποιε είναι οι επιπτώσει αυτή τη συμφωνίας για την Τουρκία. Επίση έχουμε δει μια πάρα πολύ ε, σκληρή στάση της Τουρκίας εναντίον των γυναικών και με νομοθετικό ε, ακόμα χαρακτήρα θέλουμε να ξέρουμε την σας για το θέμα αυτό. Κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ντεμιρτάς, αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια ήπια γενοκτονία σε βάρος του κουρδικού λαού ε, και ε, όπως μας είπατε υπάρχουν 500.000 πρόσφυγες, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς είναι περισσότεροι, υπάρχουν χιλιάδες νεκροί, Υπάρχει μια συνεχής δίωξη του κουρδικού λαού που αποτελεί το 25% περίπου του πληθυσμού της Τουρκίας. Είστε ικανοποιημένος από την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ανεκτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία και το καθεστώς του Ερτοάν και τη μη λήψη μέτρων και κυρώσεων εναντίον αυτού του καθεστώτος που καταδυναστεύει τον ίδιο του το λαό. Το ένα ερώτημα μου είναι αυτό. Και το δεύτερο, εσείς που είστε το 25% του πληθυσμού της Τουρκίας, πιστεύετε ότι η Τουρκία θα δεχόταν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με τον κουρδικό λαό, μιας και είστε περίπου κατοικείτε σε μια ομοιογενή περιοχή, αν εξαιρέσουμε τους Κούρδους της Κωνσταντινούπολης. Θα το δεχόταν η Τουρκία αυτό, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. please. Κύριε Τεμερτάς, παρακολουθώ τι γίνεται στην Τουρκία τον τελευταίο καιρό και πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπατε, όχι με όλα. Για τα δικαιώματα των Κούρδων πιστεύω ότι έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, διότι οι Κούρδοι μπορούν να μιλούν στις προεκλογικές εκστρατείες σε κάτι που πριν από 15 χρόνια ήταν αδιανόητο. Και είναι αδιανόητο ακόμα και σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει επίσης μεγάλες επενδύσεις υπέρ των Κούρδων. Τι έχει συμβεί, κύριε Τεμετάρς. Θέλω να σας ρωτήσω. Το κόμμα σας πότε θα γίνει ένα κοσμικό κόμμα το οποίο θα υποστηρίζει τις εθνικές μειονότητες. Είμαι από τη Βουλγαρία, στηρίζω τα μέλη της εθνικής μειονότητας, αλλά το κάνω ως ένα κοσμικό κόμμα. Καλωσορίζω κύριε Ντεμιρτάς. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή και για μας αλλά κυρίως για σας. Για μας να έχουμε μπροστά μας έναν εκπρόσωπο ενός μεγάλου κόμματος μιας χώρας που αιτείται την ένταξή της στο Κοινοβούλιο ο οποίος την επόμενη εβδομάδα, όπως ο ίδιος έχετε πει, πιθανόν να βρίσκεται στη φυλακή. Και σε εσά βεβαίω για λόγους προφανείς. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Κοινοβούλιο <clears throat> θα συνεχίσει να εργάζεται υπέρ της πράσπισης των δικαιωμάτων σας. Όμως θέλω να σας πω κάτι που μπορεί να σας απογοητεύσει. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι αρκετό. Η δύναμη των βουλευτών είναι αυτή που είναι, αλλά νομίζω ότι δεν επιδρά καθόλου πάνω στην πολιτική του κυρίου Ερτογάν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας με την σχέση αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σπρώξει τα πράγματα ένεκεν αυτή τη σχέση υπέρ τη άμβλυνση των προβλημάτων σα τουλάχιστον. Θέλω να υποβάλω και εγώ μια ερώτηση προ τη γραμμή τη ερώτηση που υπέβαλε η κυρία Πύρη. Επειδή πολλοί λένε ότι ε, πρέπει με κάποιο τρόπο να μειωθεί η παρέμβαση του ΠΚΚ, θέλω να ξέρω την άποψή σα ε, προ αυτή την κατεύθυνση. Τι ακριβώ σκέφτεστε. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Lochbiller, please. Κυρία Λόχμπιλτερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματο τη Πράσινη Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, καλώ ήλθατε και σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα δίνετε να συζητήσουμε μαζί σα. Έχετε περιγράψει τι διώξει που ε, εκκρεμούν, που ε, επαπειλούνται για εσά. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτέ Κούρδοι, όπω η Λέιλα Ζανά που είχε πάρει το βραβείο Σαχάροφ στο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε κάποιε πληροφορίε για την δική της θέση και τις εκφράσεις της ε, και, που, και τους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει. Έχετε σε αυτά τα θέματα την αλληλεγγύη μας. Επίσης φαίνεται ότι μέσω της κίνησης άρσης της ε, ασυλίας των βουλευτών θα, δεν θα, οι θέσεις οι οποίες θα κενωθούν δεν θα ξαναδοθούν στο ΧΑΝΤΕΠΕ, αλλά θα γίνουν νέες εκλογές, επαναληπτικές εκλογές και υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτές οι έδρε μπορούν να περιέλθουν στο ΑΚΕΠΕ, το οποίο θα του δώσει τα, την πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο που μπορεί να οδηγήσει και σε αλλαγή του συντάγματος. Πώς βλέπετε αυτή τη δυνατότητα. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Ντεμιρτάς και τον ευχαριστώ για την ε, συζήτηση που είχαμε και θα έχουμε στη συνέχεια. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο άνθρωπο καταδικάζει απεριφράστος την ταλαιπωρία την οποία υφίσταστε. Ε, ιδιαίτερα εγώ που είμαι Έλληνα και ανήκω στο κόμμα τη Χρυσή Αυγή που έχει υποστεί ακριβώ την ίδια δίωξη με εσάς από μια υποτίθεται δημοκρατική ελληνική κυβέρνηση έχω ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε δύο ερωτήσει: Ποια είναι η θέση σα απέναντι στη στάση της Τουρκίας για την Ελλάδα και την Κύπρο και δεύτερον πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ανέχεται τέτοιου εκβιασμούς και υποκύπτει σε κάθε πίεση του κυρίου Ροντογάν θα έχει το θάρρος να υποστηρίξει με αποτελεσματικό τρόπο την, την ε, περίπτωσή σας. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε. Αντίθετα με τον προλαλήσαντα, εγώ πιστεύω ότι έχουμε την πεποίθηση ότι υπάρχει κράτος δικαίου και στην, ε, Τουρκία, και στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τις σαφείς σας δηλώσεις. Εσείς και ο Ζαν είπατε θα μείνουμε στη χώρα μας, δεν θα προσπαθήσουμε να φύγουμε, έχετε ζητήσει την αλληλεγγύη μας. Εγώ συμμερίζομαι την άποψή σας ότι υπάρχει και μια περιφερειακή διάσταση σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της ε, Συρίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει στην Τουρκία και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει σαφή μηνύματα για τα θέματα αυτά. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρξει ανταλλαγή του, των προξενικών θεωρήσεων για τους ε, πρόσφυγες. Έχουμε επίσης ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν φύγει από τις αιστείες τους και αναρωτιέμαι τι, θέλετε, τι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Δεμιρτάς. Είμαι από το ECR. Σας καλωσορίζουμε εδώ και η μαρτυρία σας σίγουρα είναι πολύ σημαντική για μας. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ της αρχής της αυτοδιάθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάντα στηρίζω τον κουρδικό λαό και θα συνεχίσω να το κάνω και στο μέλλον. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι κινδυνεύετε με φυλέκηση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πώς θα ασκήσετε την πολιτική σας ε, δράση στη συνέχεια και επιρροή. Έπειτα, τα τελευταία χρόνια έχει χειροτερέψει η κατάσταση όσον αφορά το κόμμα σας. Και αναφερθήκατε επίσης και στις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας για το 23 και 24 κεφάλαιο που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Και είπατε ότι εσείς μπορείτε να βοηθήσετε. Η Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Δημητράς. Ε, ευχαριστώ. Πάει καιρός από τότε που βρεθήκαμε στην ε, ε, τουρκική εθνοσυνέλευση και από την άρση ασυλίας ε, των βουλευτών. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, τι μεταρρυθμίσεις ιδεοδός βλέπετε εσείς για τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Τι νομίζετε ότι χρειάζεται δηλαδή για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία και τι στοιχεία πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιηθούν για να περιοριστεί η ελευθερία έκφρασης. Δεύτερον, από διάφορους ε, στην ε, Τουρκία ακούμε ισχυρισμούς ότι το προσφυγικό χρησιμοποιείται επειδή υπάρχει και μία δημογραφική ατζέντα στο μυαλό των Ιθινόντων που θα τοποθετηθούν ε, αυτοί για να επηρεάσουν τη δημογραφική κατάσταση στη χώρα. Οι ισχυρισμοί αυτοί ισχύουν. Η κυρία Βερζιά έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου κύριε Ντεμιρτάζ, να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Είμαι φίλη της Τουρκίας, είμαι φίλη των λαών της Τουρκίας. Η πολιτιστική πολυμορφία, θρησκευτική πολυμορφία, αλλά και το κοσμικό κράτος της Τουρκίας με κάνουν να είμαι φίλη όλων αυτών. Όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι υπέρ, αλλά υπό τον όρο ότι σέβεται τα κριτήρια της Κοπεχάγης και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αυτή η άρση ασυλίας η μαζική που έκανε ο Αρτογκάν, πιστεύω ότι έχει σαν αποτέλεσμα να ξεπερνά μια κόκκινη γραμμή που εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ως ευρωβουλευτές. Και όπως είπε και κάτι πήρη, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή για αυτά τα ζητήματα. Ως ε, συμπρόεδρος της ομάδας φιλίας ε, με τον τουρκικό λαό ε, πρότεινα εταιρική σχέση, διδημοποίηση κατά κάποιο τρόπο κοινοβουλίων. Και θέλω να επανέλθω λίγο και σε αυτό που ρώτησε η Μαρία Σχάκε. Δηλαδή, κύριε Τιμιρτάς, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο τρομοκρατικός νόμος πώς χρησιμοποιείται στην Τουρκία, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Σωρίσουμε τον κύριο Δεμιχτάς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από όλε τι τοποθετήσει οι οποίε έχουν γίνει στην Ολομέλεια ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών ξέρουμε τι θέλουμε σε σχέση με την Τουρκία. Θέλουμε μια Τουρκία η οποία θα είναι δημοκρατική, να σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της, να μην φημώνει την αντιπολίτευση, να σέβεται τα δικαιώματα των Κούρδων, να μην δημιουργεί προβλήματα στη Συρία, να μην συνεχίζει να κατέχει το 40% της Κύπρου. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι στην Ευρώπη, στα άλλα Ιστιτούτα, με την πολιτική της εξημέρωσης του θηρίου και χαϊδέματος του κ. Ερτογά, έχουν αυξήσει την αλαζονία του απέναντι στην ίδια την Ευρώπη και εσείς έχετε ζητήσει πρακτικά πώς μπορούμε να στηρίξουμε γιατί πέραν του θεωρητικού επίπεδου θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρακτικά να σας στηρίξει σε αυτή την πορεία. And the last speaker is τελευταίος Καταρχάς είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνετε για ειρηνική επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Θα είμαστε δίπλα σας αν υπάρξει οποιαδήποτε ε, επίθεση της σημερινής κυβέρνησης της Τουρκίας ε, σε σχέση με τον τρομονόμο. Και θέλω να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να αποτρέψουμε μια τέτοια επίθεση εναντίον σας στο επόμενο διάστημα. Θα ήθελα να ξέρω τη θέση σας για, το, για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής, Τουρκίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό, τι προβλέπετε να γίνεται στο μέτωπο της Συρίας και κλείνοντα θέλω να επισημάνω το εξή. Οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των δίκαιων ετοιμάτων του κουρδικού λαού και των δεινών που τραβάει τα τελευταία χρόνια και πολλά χρόνια πριν στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή με μια ακροδεξιά νεοναζιστική οργάνωση στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται ως ε, εγκληματική οργάνωση θεωρώ ότι είναι γραφική αλλά και προκλητική. Ευχαριστούμε κύριε Ανδρουλάκη, λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν σας είδα, συνάδελφε. Συγγνώμη. Που άργησα, λέει η κυρία Χάρμς. Άκουσα κάποιες ερωτήσεις και νομίζω ότι με την ευκαιρία θέλω να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Επιτροπής να μας εξηγήσουν, αλλά και ο κύριος Δημητάς να μπορεί να μας πει τι έχει να πει για την παρέτηση του πρέσβου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή και για την Τουρκία αλλά και για μας ήταν μια απόφαση που προκαλεί έκπληξη. Πρέπει να ευχαριστούμε, αλλά δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω, ίσως, ε, ίσως αυτό μπορεί να το συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλη συνεδρίαση. Πολλές ερωτήσεις έχουμε κύριε Ντεμιρτάς. Ε, για τον καθένα ένα λεπτό δώστε, ίσως σε δέκα λεπτά μπορείτε να απαντήσετε όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις για σας, για το κόμμα σας, για το κράτος δικαίου, για το προσφυγικό, την τρομοκρατία, ε, τον κουρδικό λαό. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ας τελειώσουμε, αν γίνεται, στις μία παρέκκληση. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Ντεμιρτάς. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σε τόσο σύντομο χρόνο. Η κατάσταση στο Κουρδιστάν είναι πολύ σοβαρή. Δεκαετία του 90 το τοπίο ήταν παρόμοιο. Και είχαμε περίπου 3.000 χωριά και οικισμούς που έπρεπε να εκκοινωθούν. Και πάνω από 2 εκατομμύρια Κούρδοι έπρεπε να μετακινηθούν προς το δυτικό τμήμα της χώρας και σήμερα έχουμε περίπου 500.000 οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας. Οπότε δεν έχει μείνει τίποτα από τα σπίτια τους λόγω των βομβαρδισμών του πυροβολικού, λόγω των πυρκαγιών έχουν καταστραφεί τα χωριά μας. σε κάποιες πόλεις ε, έχουν σκάψει κάποια χαρακόμματα και τότε έχουμε και την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας και έχουμε αυτή την συνάδελφο, την κυρία Λέιλα, η οποία τρεις μήνες ε, βρισκόταν εκεί στο χωριό της και δεν μπόρεσε συνάδελφος να κυκλοφορήσει στους δρόμους της πόλης της επί πέντε μέρες. Το Μουσάκα επίσης έχουμε πληθυσμό πάνω από 100.000 και εκεί ε, επιβλήθηκαν μέτρα βόρειας κυκλοφορίας, καταστράφηκαν ε, σπίτια από το πυροβολικό ε, και από τα άρματα και ο κόσμος δεν μπορούσε να γυρίσει στο σπίτι του. Κατά κάποιο τρόπο έχουν τιμωρηθεί όλοι οι πολίτες της χώρας. Εκεί όμως πήραμε 90% των ψήφων ως ε, Οπότε και εμείς επιμένουμε. Θα πρέπει να μπορέσει ο κόσμος να γυρίσει στα χωριά του και θα πρέπει όλες αυτές οι ζημιές να σταματήσουν να προκαλούνται. Όμως δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση και συνεχίζουν να πλήσουν τον κόσμο που ζει σε αυτά τα μέρη. Γιατί θέλουν να σκορπίσουν τους ψηφοφόρους μας. Θέλουν έτσι να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο και την ισορροπία δυνάμεων, ιδίω εν ώψη των ε, ε, κοινοτικών, τοπικών, δημοτικών εκλογών. Να τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Όπως είπε η κυρία Πύρη, εμείς είμαστε κάθετα εναντίον χρήσης της βίας και τρομοκρατικών ενεργειών. Εμείς δίνουμε τον αγώνα μας ειρηνικά, δημοκρατικά και αυτό προτείνουμε να κάνουν όλοι οι Κούρδοι. Τα ίδια λέμε και προς το ΠΚΚ. Θα πρέπει να σταματήσει η χρήση όπλων, να σταματήσουν οι ενοπλές συγκρούσεις. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η λύση δεν δίνεται με όπλα και με τη χρήση βίας. Στη λύση θα οδηγηθούμε μόνο με διαπραγματεύσεις. Έδωσα μια σύνδεξη την περασμένη εβδομάδα και αυτό που τους είπα, να σας το επαναλάβω. Το Δεκέμβρη, πέρσι πήγαμε στο όρος Καντήλ, στο βόρειο Ιράκ και μιλήσαμε με τους ηγέτες του ΠΚΚ, εκεί στο βουνό. Θέλαμε να σταματήσουν οι όλες συγκρούσεις και αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία για να πείσουμε τους ηγέτες του ΠΚΚ εκεί και ενημερώθηκε για την κίνησή μας ο Υπουργός Εσωτερικών. Έμαθε για την επαφή μας με τους ε, ηγέτες του ΠΚΚ και ο ε, ηγέτης του, της αντιπολίτευσης το έμαθε και για αυτό του, του ε, και για αυτό και είχαμε μεγάλη δυσκολία να μπορέσουμε να κινηθούμε. Τελικά ήρθαν οι ηγέτες του ΠΚΚ και μετά από μια-δυο ώρες, ενώ εμείς ήμασταν εκεί και συνομιλούσαμε με τους ηγέτες του ΠΚΚ, ήρθε ο στρατός. Ήρθε ο στρατός και αρχίσαμε να βαλόμεθα από το πυροβολικό. Ενώ ο στρατός είχε ενημερωθεί για το ότι βρισκόμουν εκεί στο βουνό. Οπότε όταν επέστρεψα στη χώρα, όταν επέστρεψα στην Τουρκία, είπα ότι θα πρέπει τα αντιμεχόμενα μέρη να γυρίσουν τα πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και να υπάρξει κάποια αυτονομία και ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει και ότι αυτά είπαμε στο ΠΚΚ και το ΠΚΚ δέχθηκε θετικά ε, αυτές μας τις εκκλήσεις και είπαν ότι το βλέπουν θετικά να γυρίσουν στις διαπραγματεύσεις και είπαμε ότι θα πρέπει να κλείσουν αυτά τα χαρακόμματα, τα οδοφράγματα, να γκρεμιστούν που έχουν γεμίσει τις πόλεις, γιατί έχει δικαιώματα ο κουρδικός λαός. Τα ξέρουμε και αυτά επερασπιζόμαστε. Δεν χρειάζεται χρήση όπλων. Αυτά είπαμε. Και ξεκίνησε έρευνα. Όμως διατυπώθηκαν κατηγορίες εσχάτης προδοσίας. Γι' αυτό με κάτι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και έτσι δημιουργήθηκε ο φάκελος ε, της έρευνας εναντίον μου. Όλες μας οι προσπάθειες πέσαν στο κενό. Και μας είπαν οι γέρες του ΠΚΚ, καλώς, εσείς μας ζητάτε να καταθέσουμε τα όπλα, αλλά τίποτα δεν μπορείτε να καταφέρετε εσείς με την πολιτική. Το πρόβλημα δεν είναι το τι κάνουμε εμείς. Είναι η νοοτροπία του Ερντοάν και της κυβέρνησης της Άγκυρας. Αυτά είπε το ΠΚΚ. Φυσικά και εμείς βέβαια δεν πρόκειται να κατεβάσουμε τα χέρια. Θα συνεχίσουμε τις ε, προσπάθειες για να σταματήσει η χρήση των όπλων, να σταματήσει το ΠΚΚ τη χρήση ε, της βίας, αλλά και να σταματήσει και η κυβέρνηση την χρήση του στρατού. Οπότε, τι γίνεται τώρα σε όλες τις συναντήσεις μας, με το Κοινοβούλιο είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή επιτροπή. Μια κοινή επιτροπή για να εξεταστεί η υπόθεση της ειρήνευσης της χώρας. Ίσως όλες οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή επιτροπή και θα, θα πρέπει να δούμε το πώς θα επανεκκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Να υπάρξει κάποια διαμεσολάβηση, ίσως θα πρέπει να ασκηθεί πίεση προς όλα τα κόμματα ε, ούτως ώστε να επηρεαστεί και η κυβέρνηση και το ΠΚΚ. Αυτή η κοινή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει αυτή την αρμοδιότητα επισήμω. Είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι θέμα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, γιατί όταν πριτανεύει η αστάθεια, αυτό είναι αρνητικό για όλη την ε, ε, Ευρώπη. Και έγινε επομένω η επίσκεψη από την Επιτροπή του Κοινοβουλίου στις φυλακές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαπιστώθηκε ότι αυτό είναι ένα προβληματικό μέτωπο, άρα θα πρέπει να αναλάβει το Κοινοβούλιο αυτή την πρωτοβουλία. Και επί Πρωθυπουργού Νταβούτογλου αυτός ήταν ε, διαμεσολαβητής ε, με τις Φιλιππίνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κλείσαμε μια συμφωνία και ο Νταβούτογλου ήταν ο διαμεσολαβητής. Επομένως μπορεί παρόμοια πρωτοβουλία να λάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι να παρέμβει για τη λύση του προβλήματος. Σημαντικό αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουμε όσους δίνουν τη μάχη για την ειρήνη. Πανεπιστημιακοί, ε, διανοούμενοι, ε, δημοσιογράφοι, όλοι όλοι θέλουν την ε, ειρήνη. Και όλοι ανταποκρίνονται όταν αναλαμβάνει παρόμοιες πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βεβαίω αυτό θα εξωθήσει και το ΠΚΚ να σταματήσει τις ένοπλες συγκρούσεις. Τελικά θα στριμωχτεί ο Ερντογάν όσον αφορά την ανάληψη πολεμικών ενεργειών σταματήσει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Θα είναι μια ευκαιρία για μας να δώσουμε νέα όθεση, επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Και επίση αυτό θα βοηθήσει το να γίνουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Θα πρέπει να αδυνατήσει και η θέση του Ερντογάν πλευράς πολιτικής θέλει να συνεχίσει τις συγκρούσεις και τον πόλεμο, αλλά εάν φρενάρουμε αυτή την ε, τακτική, τότε θα αποδυναμωθεί ο Ερντογάν. Άκουσα τις ερωτήσεις που ήταν πολλές, μα αν ήταν τόσο εύκολο θα είχε σταματήσει το ΠΚΚ να χρησιμοποιεί τα όπλα. Αν εγώ ήμουν στο ΠΚΚ θα είχα σταματήσει τη χρήση της βίας. Εγώ κάνω τις προτάσεις μου, τις συστάσεις μου προς το ΠΚΚ, αλλά Νομίζω ότι έτσι όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, απομονωμένα δεν μπορεί να προκύψει κάποια λύση ειρήνευσης. Ε, επίσης υπάρχει και το θέμα της συμφωνίας για το προσφυγικό. Ε, εάν συνεχιστεί η αστάθεια στη χώρα θα συνεχίσουν οι πρόσφυγες να φεύγουν από την Τουρκία. Και ο πρόεδρος Ερντογάν χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως ένα δυνατό χαρτί και επιχείρημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ατού στις διαπραγματεύσεις είναι γι' αυτόν κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να εκτοπίσει και τους Αλαβίτες. Ναι, έχουμε γύρω στα 2 εκατομμύρια πρόσφυγες οι οποίοι δεν ξέρω, δεν είναι ε, προσωρινοί στη χώρα μας. Θα μείνουνε. Ήδη είναι περίπλοκε οι σχέσει. η κατάσταση. Έχουμε τους του Τουρκομάνους, Άραβες. Ήδη αυτοί είναι στη χώρα. Προέρχονται όλοι από την Συρία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί τους. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το κατά πόσον αυτή είναι οικονομικό βάρος για τη χώρα. 40% της τουρκικής οικονομίας είναι μαύρη οικονομία και είναι θέμα και οικονομικό το τι γίνεται με όλο αυτόν τον κόσμο. Αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα μείνουν ή αν θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Είναι και θέμα αν θα τους δοθεί ηθαγένεια. Πρόκειται για μια μεγάλη κρίση. Για μας είναι μια τραγωδία. Γύρω στις 300.000 Κούρδων έχουν έρθει από τη Συρία. Τους ανοίξαμε την πόρτα του σπιτιού μας. Και άρχισαν κάποιοι να επιστρέφουν στο Σαγκάλ στη Βόρεια Συρία. Κάποιοι άλλοι πήγαν στην Ευρώπη. Και αυτοί που θέλουν τη Συρία για να επιστρέψουν θα πρέπει να επανέλθει στη Συρία η ειρήνη. Θα πρέπει, η άγγελα, θα πρέπει η Τουρκία να βοηθήσει την ενευτική διαδικασία. Δεν θα πρέπει η άγγελα να βοηθά το Ισλαμικό κράτος ή την Μπόκο Χαράμ ή την Αλ Νούσρα και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Η βοήθεια που δίνεται από την Τουρκία ίσως δεν ε, γίνεται όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά αυτές όλες οι οργανώσεις δρούν στην ε, Συρία και μπορούν και δρούν ακριβώς λόγω της τουρκικής βοήθειας, της βοήθειας της κυβέρνησής μας. Και η υπηρεσία πληροφοριών MIT είδατε ότι ε, τους έδωσε με φορτηγά ε, πολεμοφόδια. Και αυτά τα φορτηγά περάσανε από τα σύνορα με την Σύρια και αυτοί οι δημοσιογράφοι που απεκάλυψαν ε, τα όσα έγιναν φυλακίστηκαν. Επομένως όταν μιλάμε για την ειρήνη να μην ξεχνούμε ότι το κουρδικό θα πρέπει να επιληθεί, θα πρέπει να ε, υλοποιηθεί πλήρως η Συμφωνία Επανεισδοχής και όλα αυτά θα καταλήξουν σε περισσότερη ασφάλεια στην Συρία. Δεν είμαστε αδύναμη χώρα, δεν μας λείπουν τα μέσα. Ο Ερντοάν μπόρεσε να επιβάλλει το καθεστώς του στην ε, Τουρκία, αλλά θα ήρθε και θα παρέλθει. Βασίζεται στην επιβολή της ε, ισχύω, βασίζεται στη στο σύγκρουση, ε, υπάρχουν τα θέματα των μειονοτήτων, Κούρδων, Αλαουιτών κλπ. Όμως εμείς είμαστε ένα απόσπαστο τμήμα του τουρκικού λαού και της χώρας. Θα πρέπει να διδρύσουμε ζωντανές τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είσαστε επικριτικοί προς τον Ερντογάν, να είστε τολμηροί. Χρειάζεται ο Ερντογάν την Τουρκία, όχι η Ευρώπη τον Ερντογάν. Γιατί 60-70% του τουρκικού λαού παραμένουν φιλοευρωπαίοι. Θέλουν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Τώρα, άλλες ερωτήσεις για τη Λέλα Οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση δεν θα πρέπει να σταματήσουν. Είπαμε για, για την απελευθέρωσή μας, είπαμε για την απαλλαγή μας. Ε, θέλουμε μια αφορμή την δίωξή μας να υπάρξει περισσότερος εκδημοκρατισμός. Το να μα πετάξουν έξω από το κοινοβούλιο βέβαια θα πάρει κάποιο χρόνο, θα πρέπει να γίνει ποινική δίωξη, να γίνει δίκη, θα πρέπει να ε, καταδικαστούμε και θα πρέπει και αυτό να περάσει και από το εφετείο και τα ανώτερα δικαστήρια. Θα πάρει χρόνο αυτό. Αλλά το εν πέμπτον των ε, βουλευτών, εάν βγουν από το κοινοβούλιο, εάν διεχθούν από το κοινοβούλιο, ε, τότε πρέπει να γίνουν πρόορε εκλογέ. Οπότε και το ΑΚΠ ε, μάλλον θα πάρει την πλειοψηφία. Υπάρχει και αυτός ο δρομοκρατικός ε, νόμος. Ε, βέβαια, ακόμα και αν καταργηθεί ο νόμος, δεν θα λυθούν τα προβλήματα, γιατί υπάρχει και ο ποινικό κώδικας που και αυτός είναι κατασταλτικός. Υπάρχουν ε, διατάξεις που φημώνουν τον τύπο, την ελευθερία έκφρασης κλπ. Όμως θα πρέπει να καταργηθούν αυτά τα άρθρα του ΠΚ. Ακόμα πάντως διατηρούμε και τις ελπίδες που συνήθως η πιο σκοτεινή ώρα είναι λίγο πριν την ανατολή του ήλιου. Δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεμίρτας. Κάνατε σχεδόν το, το αδύνατο με όλα αυτά τα ερωτήματα που σας υπευλήθησαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, ε, τις απαντήσεις σας και η ανάλυση σας ήταν πάρα πολύ σαφή. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας να ενισχύσετε το κράτος δικαίου στην Τουρκία και μπορούμε τώρα να κλείσουμε τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς που μας έδωσαν